May I Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να γυρίσετε στις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε ε, το κομμάτι της συνάντησης που αναφέρεται στο ευρώ. Κύριε Γιάννη, παρακαλώ. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Μεγάλη τιμή που μπορώ να συνομιλήσω με σας και να μοιραστώ μας με τον κύριο Γουαλτιέρη την ε, καθοδήγηση των εργασιών αυτής της συνεδρίας. Αγαπητοί φίλοι, έχω μερικά λόγια να σας πω που μπορούν να αποτελέσουν μια πλατφόρμα για τις σημερινέ μας συζητήσεις. Η διακοινοβουλευτική διάσκεψη λοιπόν στην τωρινή συνεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 20 ετία του ευρώ. Είμαστε ιδιαίτερο ευγνώμονε στου ε, εξωτερικού ομιλητές παράγοντες σημαντικού ε, στη διακυβέρνηση. Ο κύριο Αντένο καταρχά, πρόεδρο τη. Ε, Ευρωομάδας, ο κύριος Ντεγκουίντος, Αντιπρόεδρος Κεντρικής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Μοσκοβισή, Επίτροπος για τα οικονομικά, δημοσιονομικά, φορολογία, τελωνία. Έχουν δεχθεί λοιπόν να μιλήσουν σε αυτό το κέριο και πολιτικά σημαντικό ζήτημα σε αυτό το κομμάτι της συνεδρίασής μας και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με λίγα λόγια για τα πρακτικά ζητήματα. Πριν δώσω το λόγο εγώ στους ομιλητές μας, θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας περιγράψω τις διατυπώσεις για να λάβει κανείς το λόγο. Υπογραμμίζω ότι ως ήθιστε τηρούμε στο μέγιστο δυνατό τον στόχο ε, να συμμετάσχουν ως το δυνατόν περισσότεροι ομιλητές με όλο που είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Θα έχουμε λοιπόν τις εισαγωγικέ αυτές παρεμβάσεις. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα φτάσει ο χρόνος για όλους. Και γι' αυτό θα επιμείνω να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας ε, στα 2 με 3 λεπτά που θα βλέπετε άλλωστε και στις οθόνες μας να μετράνε το χρόνο. Για να μην χρειαστεί να τον περιορίσω εγώ. Θα δείτε επίσης στα τραπέζια, στα έδρανά σας, κάρτες με τις οποίες μπορείτε να υποδείξετε πως θέλετε να λάβετε το λόγο. Εάν σημαίνει αυτό, ετοιμάστε αυτή την κάρτα παρακαλώ και δώστε την στους κλητήρες μας. Αυτό ισχύει και για τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπως και στους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. In general, we will try to divide speaking time according... Και εν γέννη θα προσπαθήσουμε να κατανοούμε το χρόνο ως εξής. Δύο βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων θα ε, προηγούνται ενός ευρωβουλευτή και ούτω καθεξής. Εάν χρειαστεί όμως θα πρέπει και να προσαρμόσουμε αυτό τον τρόπο παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Και τώρα επιτρέψτε μου να κάνω το γεφύρωμα μεταξύ των χθεσινών και των σημερινών συζητήσεων με επιδίωξη να καταλάβουμε όλοι μαζί τι μας περιμένει. Ακούσαμε μέχρι τώρα τη μακροοικονομική προσέγγιση. Υπάρχουν νέοι θεσμοί, νέοι γενικοί διευθυντές, υπουργοί θα λέγαμε, νέος οδικός χάρτης ή νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων κράτη-μέλη, επενδύσεις, έρευνα, καινοτομία, ανθρωπίνο δυναμικό, όλα αυτά τα ακούσαμε. Χτες έγινε λόγος για μια ενιαία αγορά. Είδαμε όμως ότι τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν ε, προβεί και σε διμερείς συμβάσεις, μπορεί να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών. Είδαμε ότι μπορεί να αυξάνει το αριθμό των υπαλλήλων, λέει ο ομιλητής, αλλά μειώνει το χρόνο τη απασχόλησης με βάση κάποιες συμβάσει ειδικού τύπου. Επίσης βλέπουμε ότι είναι δύσκολη η διαχείριση των διαδικασιών της ε, απάτης, της φοροαποφυγής, της νομοποίησης παρανόμων εσόδων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάνουμε δισεκατομμύρια. Ακούσαμε να γίνεται λόγος για ένα μηχανισμό εγγύσεων για τις τράπεζες. Σε όλα αυτά σας παρακαλώ να μας δώσετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας έτσι ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να διατυπώσουμε την υποστήριξή μας για μια νέα μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα, χωρίς να μακρηγορώ περισσότερο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη και στους ομιλητές μας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Είναι, πιστεύω, και πανηγυρική η σημερινή συζήτηση, γιατί βεβαίως θέλουμε να γιορτάσουμε την 20 αιτία του ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο πανηγυρική, είναι αντιθέτως και μια ευκαιρία ακόμα να καταγράψουμε τα επιτεύγματά μας, να διατυπώσουμε τις ανάγκες για περαιτέρω πρόοδο. Χαίρο ιδιαίτερα που έχουμε τόσο επιφανείς ομιλητές μαζί μας. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Είμαι βέβαιος πως η συζήτηση θα είναι πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Και έτσι, περνάμε στον πρώτο μιλητή, τον κύριο Μάριο Σεντένο, πρόεδρο της Ευρωομάδας, του Eurogroup δηλαδή. Με συγχωρείτε, είστε από εδώ. Κύριε Σεντένο, έχετε το λόγο. Good morning. Thank you, Chair. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων τη Ευρώπη, κύριε Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας ομιλώ σήμερα κατά την επέτειο της 20 ετίας από την εισαγωγή του ευρώ για να συζητήσουμε το μέλλον του αλλά και να καταγράψουμε τα επιτεύγματά του. Είναι η δεύτερη φορά που έχω την ευκαιρία συμμετάσχω σε αυτή την κοινοβουλευτική εβδομάδα. Μια πρωτοβουλία που εκτιμώ ιδιαίτερος και χαίρομαι που μπορώ να συμμετέχω οικονομική και νομισματική πολιτική στην Ευρώπη. Εμφανίζεται από τα πρώτα βήματα της δημιουργίας της Ευρώπης Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με το ευρώ που είναι όχι μόνο ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητας αλλά και το δεύτερο σε μέγεθος ευρωπαϊκό ε, παγκοσμίως νόμισμα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείχνει ο πολίτης, πολύ περισσότερο από ότι ποτέ. Βέβαια δεν ήταν ε, το μονοπάτι αυτό που διαβήκαμε χωρίς δυσκολίες την τελευταία 20 ετία. Η κρίση έχει δοκιμάσει το ευρώ, έχει καταγράψει σφάλματα, έχει καταδείξει σχεδιαστικά λάθη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ωστόσο, με όλες τις αντικσότητες, η αποφασιστική δράση και η πολιτική έδωσαν ένα ισχυρό ευρώ. Και έτσι έχουμε ένα γυρό, γερό ε, νόμισμα, ένα αγκίστρωμα το οποίο, στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η οικονομική μας πολιτική και το μέλλον το μέλλον όπου ε, μπορεί να αμφισβητούνται πολλά από τα δεδομένα μας όπου η τεχνολογία και η καινοτομία έχει φτάσει σε ανυπέβλητα ύψη, όπου οι ανισότητες επικρατούν, όπου ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι αδυσόπιτος και όπου υπάρχει πολύ έντονος λαϊκισμός και κίνδυνη πολιτική. Χαμηλή ανεργία, υψηλή απασχόληση, αυξανόμενη μισθή και 22 αλλεπάλληλα τρίμηνα ανάπτυξης είναι φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν κάνει να καμφθεί αυτή η δυσφορία που εκφράζεται από τον κόσμο. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αιτίες αυτού του κακού. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Πιο έντονη οικονομική συνεργασία, συντονισμό μεταξύ των μελών της ε, Ευρωζώνης με 1,5% το 2017 και τη χαμηλότερη απόκληση στις οικονομικές δραστηριότητες, στις οικονομικές επιδόσεις, πάλι είναι φαινόμενα τα οποία δεν αρνούμαστε, αλλά πάλι δεν έχουν δώσει το αποτούμενο αποτέλεσμα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, πρέπει να γίνει πιο ανθεκτική, πιο συμπεριεκτική η οικονομία μας και η έννοια συμπεριεκτικός είναι πάρα πολύ απλή. Κατά μέσο όρο αναπτύσσονται οι οικονομίες μας, ναι αλλά ο μέσος όρος μπορεί να είναι απατηλός. Οι πολίτες που, έχουν, που ανήκουν στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα ή κατανομή εισοδήματο είναι όλο και περισσότεροι. Αλλά καλύπτεται αυτός ο αριθμός γιατί αυξάνεται το εισόδημα των πολύ πιο πλούσιων ολίγων και έτσι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση για τους πολλούς, όχι για τους λίγους. Αυτό σημαίνει να διανομή εισοδήματος. Πρέπει να, ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα, σε όλες τις χώρες. Στην, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι σε θέση να αντλήσει τα ωφέλη από το ενιαίο νόμισμα. Πολλά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί ήδη προς την ορθή κατεύθυνση. Έχει ξεκινήσει η Τραπεζική Ένωση, έχει εγκαθιδρυθεί ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα. έχουμε βελτιώσει το συντονισμό, την πολιτική συντονισμού. Έχουμε υιοθετήσει μια σειρά από σκληρέ μεταρρυθμίσει σε εθνικό επίπεδο, κρίσιμη δράση, κρίσιμε δράσει για να εξασφαλιστεί σταθερότητα, κρίσιμε αλλά όχι επαρκή και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη σταθερότητα. Yeah, το Eurogroup λοιπόν δουλεύει ακόμη περισσότερο για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. με δουλειά που οδήγησε στα αποτελέσματα της ε, ε, Ευρωσυνόδου Κορυφής ε, του Δεκεμβρίου και το Ταμείο, το Ταμείο Εκαθάρισης, ένα ακόμα πολύ σημαντικό βήμα δηλαδή για την Τραπεζική Ένωση, αλλά και για τα, με τα δημοσιονομικά μέσα για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα για την Ευρωζώνη. Το Eurogroup έχει λάβει εντολή να συνεργαστεί και να καταθέσει νέες και αποτελεσματικέ προτάσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Στους επόμενους τρει μήνες λοιπόν θα επικεντρωθούμε στα εξή ε, καθήκοντα. Πρώτα θα πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις τροποποίησεων για τη συνθήκη που αφορά τον Ευρωπαϊκό Σταθεροποιητικό Μηχανισμό. Δεύτερον πρέπει να κοιτάξουμε περαιτέρω βήματα τη Τραπεζική Ένωση, διασφαλίσει καταρχά και ζητήματα ρευστότητα στον ενίο μηχανισμό καθάρισης και επίσης πρέπει να βρεθούν δημοσιονομικά μέσα για την ανάπτυξη με ένα βήμα ιστορικό στην ιστορία της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι και πιστεύω πως το μέσο αυτό θα είναι ένα σημείο κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης. Επίσης, το Δεκέμβριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν την εγκαθίδρυση αυτού του μέσου επειδή ακριβώς αντελήφθησαν συλλογικά πως υπήρχε ένα κρίσιμο κενό στο νόμισμα, μια ενιαία νομισματική πολιτική πρέπει να συμπληρώνεται και από το κατάλληλο και στοχευμένο δημοσιονομικό μέσο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι πρόσθετο στα μέσα τα οποία έχουν στη θέση τους όλα τα κράτη-μέλη και που αιτιολογούνται και από τις κοινέ πολιτικές. Με άλλα λόγια, δεν μιλούμε για έναν εξοραϊσμό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ούτε και μιλάμε για τον κατακαιρματισμό σε δύο τμήματα του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου με διαφορετική γραμμή για, την, ε, για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και διαφορετική γραμμή, κονδύλια δηλαδή, για τις χώρες του ευρώ. Έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένα κριτήρια και στόχους του ευρώ και πρέπει να βελτιωθεί και η ελκυστικότητα και η αποδοτικότητα της ευρωζώνης με θετικά αποτελέσματα που θα ενθαρρύνουν τα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιταχύνουν και να βελτιώσουν τις προσπαθίες τους για ένταξη στην ευρωζώνη, προοπτικές που βεβαίως ε, θα στηρίξουμε και εμείς σε όρους τεχνικούς και δημοσιονομικού. Πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια σε δύο παράλληλους στόχου. σύγκληση αφενός, ανταγωνιστικότητα αφετέρου και επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί έχει σημασία να σταθούμε και στα δύο. Η σύγκληση στις ε, συνθήκες διαβίωσης. Είναι ένα από, τα κύρια, από τις κύριες υποσχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωποίησης για την Ευρωζώνη, όμως έχει επιπλέον μεγάλη σημασία, γιατί κάθε ε, ε, σημαντική διαφορά, οι μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών της Ευρωζώνης θα έχει σημαντικές συνέπειες στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης και η κρίση έδειξε ότι είναι πραγματικό ο κίνδυνος της διάχυσης των προβλημάτων επιπλέον. Οι θεσμικές δομές αλλά και οι επιχειρηματικοί κύκλοι των κρατών μελών, εάν γίνουν πιο ενοποιημένοι, τότε θα είναι και πιο αποτελεσματική η νομισματική ένωση, πιο ωφέλιμη δηλαδή η συμμετοχή στην ευρωζώνη. Το ίδιο ισχύει και για την ανταγωνιστικότητα. Είναι απαραίτητο για να μπορεί κάθε χώρα να αντιμετωπίσει την μεγάλε τις μεγάλες προκλήσεις παγκοσμιοποίησης και του παγκόσμιου ανταγωνισμού, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε συνάφεια με τα λοιπά κράτη της ευρωζώνης, για να μην υπάρχει η επιβράδυνση αυτή. Έτσι λοιπόν ε, είναι σαφές ότι οι χώρες της Ευρωζώνης ε, χώρε Ευρωζώνη πρέπει να έχουν υψηλότερε προδιαγραφές ανταγωνιστικότητα και σύγκληση, έχοντα πάντα αυτή την ε, κυριαρχία στην νομισματική πολιτική. Και εδώ έχουμε το δημοσιονομικό μέσο. Ε, πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς μπορεί να στηρίξει τη σύγκληση αλλά και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη αυτό το δημοσιονομικό μέσο. Γιατί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, υπάρχει μια σειρά από εργαλεία που καλύπτουν ευρύ τομεί πολιτική, ε, για το ευρώ και τις ανάγκες του. Όμως αυτά τα εργαλεία πρέπει να ξεπερνούν και να συμπληρώνουν αυτό που ήδη υφίσταται στο ΟΠΟΥΔΟΠΟΥ. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποστηριχθούν νέες μεγάλες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις για καλύτερη παραγωγικότητα, για γρήγορη αναδιανομή των πόρων ε, σε εργατικό δυναμικό αλλά και κεφάλαιο στην Ευρωζώνη Πρέπει να αντισταθμιστούν τα προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις φερρυπίν στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης και, και νόημα θα είχε επίσης και να γίνουν ιδιαίτερες επενδύσεις, κυρίως δημοσίου χαρακτήρα, για να ενισχυθεί το δυναμικό της Ευρωζώνης και το αναπτυξιακό δυναμικό γενικότερα της περιοχής της Ευρωζώνης. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να διαφυλάξουν χώρους κέριους όπως την έρευνα, την ανάπτυξη, τεχνολογία, την εκπαίδευση, τις υποδομές, ε, με σταθερές και στοχευμένες επενδύσεις μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της, του δυναμικού της οικονομίας μας, να παράγει και να προσαρμόζεται. Κάθε οικονομία δηλαδή, αλλά και το σύστημα στο συνολό του μπορεί να γίνει πολύ πιο ανθεκτική και ανθεκτικό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μόνο, σε, μόνο τις εθνικές δράσεις θα συμπληρώνει ένα τέτοιο εργαλείο, ούτε και θα απαλλάσσει τις χώρες από, από την υποχρέωση να υιοθετούν και να εφαρμόζουν υγιείς δημοσιονομικά πολιτικές. Πάντα θα πρέπει κάθε χώρα να ε, ακολουθεί και να ενστερνίζεται, αλλά και να έχει την πρωτοβουλία υγιών δημοσιονομικών ε, πρωτοβουλίων και δράσεων η πηγή χρηματοδότησης και πάνω απ' όλα το μέγεθος του μέσου αυτού που προξενούν πολλές ανησυχίες, πολλές νέες ε, ε, ιδέες ή σενάρια θα ακουστούν φαντάζομαι στους επόμενους μήνες άλλοι θα το επικρίνουν ως υπερβολικό, υπερβολικά υψηλό άλλοι ως υπερβολικά ανεπαρκές εμένα δεν με απασχολεί αυτό το ποσό δηλαδή το χρηματικό ε, δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί βεβαίως ναι μπορεί να περιορίσει το τι θα κάνουμε αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι να έχει αποτελεσματικότητα αυτό το εργαλείο, να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αξιοποίηση του, να αποδείξουμε ότι είναι ένα τρόπο αποτελεσματικό, να βάλουμε πάλι μπρο το κινητήρα τη ευρωπαϊκή οικονομία και να το προσαρμόσουμε συν το χρόνο και με την εμπειρία που θα συλλέγουμε και μακροπρόθεσμα το μέσο αυτών. Βεβαίω και θα φέρει τα αποτελέσματα που θα έχουμε σχεδιάσει και μέχρι εκεί που θα το έχουμε πάει εμεί. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, σα διαβεβαιώ διακυβέρνηση τώρα. Η διαδικασία για τη διαχείριση του μέσου δεν έχει την προσοχή που θα άξιζε συγκεντρώσει. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν και ευελιξία για να μπορεί να προσαρμόσει τις ανάγκες της Ευρωζώνης, να συνδεθεί το εργαλείο με, τον, με το Ευρωπαϊκό Εξάτμινο και τον Οικονομικό Συντονισμό. Θα πρέπει να μπορεί το Eurogroup να περιγράφει τις κύριες γραμμές βεβαίως υπό την κατεύθυνση που, καθοδήγηση που θα δώσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων με βάση κριτήρια των κρατών της Ευρωζώνης όπως άλλωστε έχει ήδη σημειωθεί. Και αυτό πρέπει να μεταγραφεί σε όρους θεσμικούς, στέρεους νομικά, με συγκεκριμένε συνέπειε και όρια ω προ τη χρηματοδότηση. Και πριν να κλείσω, σα διαβεβαιώ ότι προτίθεμαι να ολοκληρώσω. Επιτρέψτε μου δύο λόγια ακόμα να πω για τη διαδικασία. Το Eurogroup θα ετοιμάσει συμφωνία ως προς τα χαρακτηριστικά του μέσου αυτού μέχρι τον Ιούνιο για να μπει μετά στην νομοθετική διαδικασία αυτή η πρόταση. Εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ξέρω ότι ήδη έχετε ξεκινήσει τη δουλειά για τις δημοσιονομικές δυνατότητες της Ευρωζώνης εδώ και μερικά χρόνια. Περιμένω να ακούσω συγκεκριμένε προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει στη διαμόρφωση του τελικού αυτού μέσου και είμαι στη διαθεσή σας για ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. Για να ολοκληρώσω και ζητώ συγγνώμη για το ότι μακρηγόρησα και ξεπέρασα τα χρονικά όρια. Στο διάρκεια του 2019 θα δούμε πολλά πράγματα να αλλάζουν στο ευρωπαϊκό οικονομικό και δημοσιονομικό τοπίο με δεδομένη την επιβράδυνση και τους κινδύνους που διαγνώσκουμε χρειάζεται ο συντονισμό της δράσης μας. Εγώ θα σταθώ σταθερός στη στόχο των μεταρρυθμίσεων. Με αποφασιστικότητα πιστεύω θα μπορέσουμε να τις εισαγάγουμε και το εργαλείο αυτό για έναν ε, ειδικό προϋπολογισμό, μια ειδική διαχείριση δημοσιονομική της Ευρωζώνης είναι ένα σαφές μια σαφής απόδειξη της βούλησής μας, της βούλησής μας να στηρίξουμε το ευρώ, της αποφασιστικότητάς μας, αυτή η, η ιστορία του ευρώ να στεφθεί με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και στο σύνολο που Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα. Συγχαρητήρια. Πραγματικά αναφερθήκατε σε όλα τα θέματα, τα ευαίσθητα θέματα. Και υπάρχουν χρήματα και για τη σύγκληση και για την ανταγωνιστικότητα, οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι μηχανισμούς σε αυτή τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή είναι ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής. Παραμένουν ανισορροπίες, ε, παραμένουν κάποιες αδικίες, αλλά Μέρος των μηχανισμών αυτών έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Επόμενος ομιλητής μας είναι ο Λουίς ε, Κουίντος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, κύριε Επίτροπε Μασκοβισή, Πρόεδρε του Eurogroup, κύριε Σεντένο, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας που με έδωσαν την ευκαιρία να έρθω εδώ και να συζητήσω μαζί σας για τα πρώτα 20 χρόνια του ευρώ και τι μας περιμένει στη συνέχεια. Οι δύο πρώτες δεκαετίες του ευρώ ήταν ε, πραγματικά εξαιρετικές, διότι αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση που οδήγησε σε απώλειες βέβαια για όλες τις οικονομίες ολόκληρο το κόσμο και επίσης αντιμετώπισε και την δημοσιονομική κρίση που απέλησε το ίδιο το ενίο νόμισμα. Έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση προχώρησε σε δύο στάδια. Όμως η ολοκλήρωση πλήρης της ΟΝΕ σημαίνει ότι όταν έχουμε τέτοιες ε, ταραχές η σύγκληση που είχαμε πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό δυστυχώς δεν μπόρεσε να προχωρήσει αντίθετα έκανε ε, βήματα πίσω. Βρεθήκαμε σε μη υπαρξιακή κρίση. Χρειάστηκε ε, μια διόρθωση. Οι ανισορροπίες όντως διορθώθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό, οι ανισορροπίες ευελτιώθηκαν και τα δημοσιονομικά ελλείμματα μειώθηκαν. Σαν αποτέλεσμα και χάρη και στη στήριξη της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρωζώνη ε, μπόρεσε να μπει σε πορεία ανάπτυξη που οδήγησε σε βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασία και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο χώρος εδώ μας επιτρέπει να συζητήσουμε και τον ρόλο των κοινοβουλίων στο ταξίδι αυτό. Τα κοινοβούλια έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε παραπάνω και να συνεισφέρουμε στη βελτίωση της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η Ένωσή μας, όπως ξέρετε, βασίζεται στην αξία της δημοκρατίας και στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και τις παραδόσεις που βασίζονται σε μηχανισμούς και θεσμούς που προστατεύουν την ελευθερία, τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και είναι κατά βέβαια κάθε κατάχρηση εξουσίας. Η νομιμότητα λοιπόν σε ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε, ο Δήμο μα δηλαδή, να έχουν την επιλογή και να έχουν και φωνή. Από την άλλη βασίζεται και σε θεμελιώδεις κανόνε που αποτελούν και τη βάση του κοινωνικού μα ε, συμβολέου. Οπότε η νομιμότητα από μόνη της δεν φτάνει. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια από τους θεσμούς. Θα σας δώσω παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει δημοκρατική εντολή ε, που αναφέρεται στις συνθήκες και έχει επικυρωθεί από όλες τις χώρες μέλη βάσει των συνταγματικών τους διαδικασιών. Στην εντολή αυτή λοιπόν και για να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους μηχανισμούς εφόσον είναι αναγκαίο. Και η ανεξαρτησία της προστατεύεται και η νομιμότητα των αποφάσεώς της δεν υπονομεύεται από πολιτική ανάπτυξη ή για λόγους βραχυπρόθεσμου εκλογικού κέρδους. Ε, το, από την άλλη μεριά, εκτό από την εξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει λογοδοσία προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί του λόγου τη Ευρώπη. Και αυτό συμπληρώνεται και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από την αποτελεσματικότητα, ε, η αποτελεσματικότητα επίση στη διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυσφαλίζεται από το Ελεκτικό Συνέδριο. Και όλα αυτά για να τηρούμε την εντολή μα και να μην ε, δρούμε αυθαίρετα. Λογοδοτούμε λοιπόν πολύ σοβαρά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύξει μια, ένα πλαίσιο λογοδοσίας που πηγαίνει πέρα από τις απαιτήσει της συνθήκης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά τακτικά και σε βάθος μας ελέγχει όπως θα έπρεπε και όπως περιμένουμε κατά τη διάρκεια της κρίσης ο έλεγχος αυτός ανέβηκε σε κλίμακα. Τώρα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αυτούς τους συγκεκριμένους κανόνες. Εμείς προσπαθούμε να ε, βελτιώσουμε την νομιμότητα και οι θεσμοί να λειτουργούν όσο γίνεται καλύτερα και να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικέ. Σε αυτέ τι ζητήσει συζητάμε για το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα και τη λογοδοσία. Και αυτό είναι αλήθεια κυρίως για αποφάσεις που έχουν να κάνουν με οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα, τα οποία είναι και ιδιαίτερα πολιτικά. Επ' αυτού λοιπόν και τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη αναλάβει σημαντική ευθύνη. Τα Εθνικά Κοινοβούλια εγκρίνουν τον εθνικό προπολογισμό και τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Συγχρόνω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι συνομοθέτη, παίζει ένα σημαντικό ρόλο για το σχεδιασμό και την ε, αποτελεσματική χρήση του πλαισίου διακυβέρνηση. Αυτή η κοινοβουλευτική ευρωπαϊκή ομάδα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μα επιτρέπει να μάθουμε ένα από τι εμπειρίε του άλλου. Στην πραγματικότητα, Υπάρχουν πολλέ επιτυχεί μεταρρυθμίσει σε διάφορε πολιτικέ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα έρθω σε συγκεκριμένα παραδείγματα για τι δημοσιονομικέ υπηρεσίε. Η Τραπεζική Ένωση είναι πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση τη ΟΝΕ. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα από την κρίση. Έχουμε σημαντικά και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχουμε την εποπτεία των τραπεζών. Πέντε χρόνια τώρα, η οποία μας ε, οδήγησε να καταλήξουμε στο πόσο εποπτεύουμε και ελέγχουμε τις τράπεζες. Με ένα νέο πλαίσιο επίσης εξυγίαση, το οποίο διασφαλίζει ότι όταν έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, τότε δεν πληρώνουν οι κυβερνήσεις και ο κόσμος, αλλά ο δημοσιονομικός τομέας. Βοηθάει επίση η Τραπεζική Ένωση οι τράπεζε να είναι πιο ασφαλεί και να μπορέσουν να αντέξουν και να στηρίξουν καλύτερα την ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε πετύχει πρόοδο, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει το έργο μα. Από τη μία πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση χρησιμοποιώντας τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και να προχωρήσουν οι πολιτικές συζητήσεις για τον τρίτο πυλώνα που λείπει ακόμα στην Τραπεζική Ένωση και που είναι η εγγύηση και οι ασφαλείς καταθέσεων. Η ολοκλήρωση λοιπόν της Τραπεζικής Ένωσης προχωράει και η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί. Χρειάζεται, ε, μάλλον η πρόοδος όμως η επιπλέον εξαρτάται και από το εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει εναρμόνιση παρόλο που πολλά ζητήματα είναι στα χέρια του εθνικού νομοθέτη. Η διαιτησία, η ισοτιμία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά όμως μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ευρωπαϊκή νομοθεσία και κοινού θεσμούς που σημαίνει ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά με την άλλη. Τα Εθνικά και τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια θα πρέπει να ζουν σαν να είναι δύο που τρέχουν συγχρόνως και όλοι εξαρτώνται από την νομιμότητα. Δηλαδή πρέπει να συνεργάζονται. Η μία ομάδα πρέπει πάντα να διασφαλίζει την νομιμότητα του παιχνιδιού. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε την απόδοση ευθυνών και πώς αυτές καταμερίζονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να γίνεται από την πίσω πόρτα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη δημόσια συζήτηση. Κάθε χρόνο λοιπόν αυτή η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα μας, επιτρέπει αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λουίς Ντεγκίντο, σας συγχαρητήρια και για την επέτειο του ευρώ και για την επιτυχημένη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις κρίσεις. Καταλάβαμε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ταμείου εξασφάλισης είναι για τις ε, αποταμιεύσεις και τις καταθέσεις είναι αυτό που ζητάει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω όλε οι μεταρρυθμίσει, αγαπητοί συνάδελφοι, όλα τα εργαλεία βρίσκονται στα χέρια ενό και μόνο ατόμου, δηλαδή του αρμοδίου επιτρόπου, του κυρίου Πιάχ Μοσκοβισή, του επιτρόπου αρμοδίου, αρμοδίου για την φορολογία, για τα τελωνία, για τα χρηματοπιστωτικά. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπερβάλλετε λίγο για τι αρμοδιότητε και την έκταση του χαρτοφυλακίου των υποχρεώσεων μου, αλλά με χαρά θα σταθώ στο ύψο της ε, Κύριε Σεντένο, κύριε Ντεγκίντο, αγαπητοί βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, καλημέρα σε όλου. Πράγματι, είπε ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη ότι σήμερα είναι μέρα εορτασμού τη 20 η επαιτίου του ευρώ και είμαι εδώ μαζί σα για να το γιορτάσουμε μαζί. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να εκτιμήσουμε τη διαδρομή που έχει διανύσει το δικό μα ενίο νόμισμα τι τελευταίε δεκαετίε, τι δύο τελευταίε δεκαετίε, την επιτυχία του, τα εμπόδια που κατάφερε να υπερπηδήσει και τι προσπάθειε που θα πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε να καταβάλουμε για την οικονομική και νομισματική ένωση. Το ευρώ είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο απτά ευρωπαϊκά επιτεύγματα. 360 εκατομμύρια πολίτες περίπου και σχεδόν χρησιμοποιούν ένα νόμισμα, γνωρίζουν για ένα νόμισμα ε, το οποίο ανήκει σε όλους μας. Είναι εξαιρετικά δημοφιλές το 74% των πολιτών θεωρούν ότι ωφελεί την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση και όσοι ονειρεύονται να φύγουν από το ευρώ και ε, ε, τροφοδοτούν το λαϊκισμό τελικά διαψεύδονται, αποδεικνύεται αυτό ότι διαψεύδονται ξανά και ξανά. Είναι μια ισχυρή εμπορική και οικονομική δύναμη στο κόσμο. Είναι το δεύτερο διεθνές νόμισμα. Περίπου 60 χώρες χρησιμοποιούν ή θα αρχίσουν να το χρησιμοποιούν λίαν συντόμως. Είναι οι καλύτερες επιδόσεις από, ε, από οποιαδήποτε επίδοση είχε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό εθνικό νόμισμα στο παρελθόν. Όμως ε, τέθηκε σε κίνδυνο και δοκιμάστηκε η στεναρότητα του νομίσματός μας. Η κρίση του 2018 και 2015-2018 απόδειξε ε, τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ευρώ και μπροστά στον κίνδυνο που βάρινε το σύνολο της ζώνης του ευρώ, το ενιαίο νόμισμα απέδειξε ότι είναι ανθεκτικό. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν έλαβαν ισχυρέ αποφάσει, τα κράτη-μέλη έλαβαν ισχυρέ αποφάσει για να ενισχύσουν την ΟΝΕ. Έγιναν θεσμικέ αλλαγέ. Μιλώ για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, στον οποίο θα αναφερθώ και αργότερα. Ενισχύσαμε το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών και δημοσιονομικών μα πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και σήμερα λοιπόν τα αποτελέσματα είναι εδώ, απτά μπροστά μα. Έχουμε αφήσει την οικονομική κρίση πίσω μα, οριστικά κιόλα. Και ε, η ανακοίνωση τη Επιτροπή αποδεικνύει ότι η ανάκαμψη υπάρχει και η ανάπτυξη έχει επιστρέψει παρόλο που ελοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι και υπάρχουν κάποια σύννεφα. Η αγορά της εργασίας βελτιώνεται σημαντικά σε όλες τις χώρες. Επομένως το νέο νόμισμα έχει βγει ενισχυμένο από αυτή την κρίση. Ο συνάδελφος Μάριος Σεντένο μας μίλησε για αυτή την οικονομική κρίση η οποία μας έκανε να περάσουμε σε πολιτική κρίση. Όξυνση και αύξηση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των χωρών της ζώνης του ευρώ και από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό περιπλέκει την καθοδήγηση της οικονομικής πολιτικής διότι υπάρχει θεμητό το αίσθημα της αδικίας που τροφοδοτεί τον ευρωσκεπτικισμό και πρέπει να ανταποκριθούμε και να απαντήσουμε σε, αυτή τις ερωτήσεις και να μειώσουμε τις ανισότητες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεταρρυθμίσεις που να ενισχύουν τη σύγκληση μεταξύ των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και που ενισχύουν τη δυνατότητα σταθεροποίησης και αντοχής, ανθεκτικότητας του ενιαίου νομίσματος. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σκόλπο του Eurogroup ε, έκανε την εμβάθυνση της ζώνης του ευρώ προτεραιότητά της και θέλω να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για τη στήριξη που έχουν δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά τα χρόνια. Επιδιώκουμε προτεραιότητες. Πρώτον, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Πολλά ήδη έχουν γίνει με την οικονομική κρίση. Έχουμε ένα μηχανισμό ενιαίο ε, ε, εποπτείας των τραπεζών, ταμείο για την εξυγίαση των τραπεζών, ε, όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί τα καθήκοντά μας. Έχουμε προόδους που πρέπει ακόμα να σημειώσουμε, πρέπει ακόμα να επιτύχουμε. Ε, στην τελευταία σύνοδο της ζώνης του ευρώ έγιναν πολύ σημαντικές εξελίξεις. Συμφώνησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη δημιουργία ενός δικτυού ασφαλείας για ένα ενιαίο ταμείο για την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, κάτι πολύ σημαντικό για την τραπεζική ολοκλήρωση, για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Συμφώνησαν επίσης οι ηγέτες ότι ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητα θα ε, προσφέρει στήριξη και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Ωστόσο, λείπει ο τρίτος πυλώνας από την Τραπεζική Ένωση, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων, των τραπεζικών καταθέσεων και αποταμιεύσεων δεν ε, είχαμε μιλήσει μόνο για την εποπτεία και επιθεώρηση, δεν είχαμε μιλήσει μόνο για την εξυγίαση, αλλά και για την εγγύηση των καταθέσεων. Είναι μια συμφωνία που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα μεταξύ κρατών μελών. Λυπούμε γιατί δεν έχει γίνει η απαραίτητη πολιτική πρόοδο σε αυτό το επίπεδο. Ήδη το Δεκέμβριο μειώσαμε πάρα πολύ το κίνδυνο, άρα πρέπει να μάθουμε να τον μοιραζόμαστε αυτόν τον τόσο μειωμένο κίνδυνο. Δεύτερο πυλώνα, η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Χαίρομαι για τι πρόοδου που έχουν σημειώσει τα κράτη-μέλη. Έχουμε τη συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ασφάλειας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανση των Τραπεζών. Είναι μια εργαλειοθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για να προστατεύονται καλύτερα τα κράτη-μέλη ε, ε, από τη στιγμή που τα θεμελιώδη οικονομικά του στοιχεία είναι ισχυρά σε περιόδου κρίση. Θα πρέπει ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα να μεταρρυθμιστεί έτσι περαιτέρω, κατά την άποψή μου. Και για να μιλήσω με ειλικρίνεια, γιατί γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, είναι δύσκολα αποδεκτό ένα όργανο που παίρνει τόσο δεσμευτικέ αποφάσει να απαλλάσσεται από κοινοβουλευτικό έλεγχο στέρεο και στεναρό. Να είναι ένα όργανο αμυγό διακυβερνητικό. Είναι δύσκολα αποδεκτό κάτι τέτοιο, όπω λέω. Και γι' αυτό προτείνουμε να θεσπιστεί ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητας ε, στο ευρωπαϊκό νομοθετικό κεκτημένο να γίνει το ευρωπαϊκό νομισματικό Δημοκρατικό Ταμείο να έχει έναν Υπουργό Οικονομικών, ο οποίο δημοκρατικό να ορίζεται και να είναι υπόλογο και υπεύθυνο έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο και θα παντά. Και χαιρετίζω την ποιότητα των κοινοβουλευτικών σα εργασιών ε, με αυτό το θέμα. Τρίτη προτεραιότητα είναι αυτό που ανέφερε ο Μάριο Σεντένο. Ε, ε, δημιουργία ενό. Ε, δημοσιονομικού εργαλείου για τη ζώνη του ευρώ, περιοπολογισμού δηλαδή, για να ενισχυθεί η σύγκληση εντό τη ζώνη του ευρώ με στόχο την μείωση των αποκλήσεων, των ανισοτήτων που υπονομεύουν την συνοχή μα. Και εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε δύο φιλόδοξε προτάσει για την περίοδο 2021-2027, γιατί έχουμε συγκλίνει τι απόψει μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και πιστεύουμε ότι ο προπολογισμό τη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρο του κοινοτικού προπολογισμού αυτού καθεαυτού. Να μην ξεχνούμε αυτό το εργαλείο σταθεροποίησης και αλληλεγγύης που θα προστατεύει τις δημόσιες επενδύσεις σε περίπτωση μεγάλων ασύμετρων σοκ στην οικονομία. Ε, έτσι θα μετριάζεται ο αρνητικός αντίκτυπος των μεγάλων ασύμετρων σοκ και θα έχουμε ενίσχυση ε, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Οι Υπουργοί Οικονομικών λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουν στα χαρακτηριστικά αυτού του μηχανισμού που θα βοηθάει τη σύγκληση και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ. Σήμερα συνεχίζουμε συνεχίζονται οι συζητήσεις εντός του Eurogroup ε, και θα συνεχιστούν μέχρι και τον Ιούνιο. Έχουμε λοιπόν μια συμφωνία επί τη αρχής για το εργαλείο αυτό, αλλά απέχουμε πολύ από τι πρακτικέ λεπτομέρειε εφαρμογή από συμφωνία επ' αυτών. Ελπίζω ότι θα συμμετάσχει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη εβδομάδα, στον Σύνοδο του Ιωνίου, ε, την πρώτη εβδομάδα και ότι μέχρι τότε θα έχουμε πολύ σημαντική πρόοδο. Εμεί θα εργαστούμε με όλε μας τι δυνάμεις. Χρειαζόμαστε αληθινό προπολογισμό εξοπλισμό της ζώνης του ευρώ. Γιατί θα λειτουργήσει και σταθεροποιητικά σε βάθος χρόνου. Η ισχύς η δυνατότητα ελιγμών, η δυνατότητα χειρισμών για τη ζώνη του ευρώ είναι καθοριστικοί παράγοντες και θα γίνουν και θα μπορέσουμε να τους εγγυηθούμε με τον προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα της διακυβέρνησης. Υπάρχει δημοκρατική απέτηση, απέτηση για εκδημοκρατισμό ε, γι' αυτό θα συνεχίσω να συνηγορώ υπέρ της ύπαρξης θέσης Υπουργού Οικονομικών της Ζώνης του Ευρώ που θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα προεδρεύει του Συμβουλίου το οποίο θα ονομάζεται Eurogroup αλλά το οποίο θα είναι επίσημο Συμβούλιο Υπουργών και δεν θα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που να μην υπόκεινται σε έλεγχο του Κοινοβουλίου. Και πρέπει να αυξήσουμε το διεθνή ρόλο του ευρώ, να τον ενισχύσουμε. Έχουμε εξοδαφικές κυρώσεις που λαμβάνονται π.χ. από τη ΣΥΠΑ και αυτό έχει αντίκτυπο σε εμάς, το υφιστάμεθα σήμερα. Ενισχύοντας λοιπόν το ρόλο του ευρώ θα μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αυτονομία στη στρατηγική μας και θα μπορούμε να υψώσουμε το ευρώ ως διεθνές νόμισμα ε, με συναλλακτική αξία εξίσου σημαντική όπως αυτή του δολαρίου. Κυρίε και κύριοι, το ευρώ είναι 20 ετών έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, μεγάλη διαδρομή. 20 χρονών όμως κανείς είναι ακόμα νέος και χρειάζεται στήριξη και γι' αυτό πρέπει να παραμένει βασική μας και απόλυτη προτεραιότητα. Πλησιάζουν οι ευρωπαϊκές εκλογές και δεν θα πρέπει να μας ε, παρασύρουν μακριά από τη δράση. Θα πρέπει οι ευρωεκλογέ να λειτουργήσουν ως ε, βελόνα στάθμισης ε, έτσι ώστε να ε, επιστρέψει, να γίνει ζυγοστάθμιση αν θέλετε και να ε, ε, έρθει στο επίκεντρο αυτό που πραγματικά μας απασχολεί, το οποίο είναι η σταθεροποίηση. Είμαι πεπισμένος ότι η στήριξη, η πολιτική πίεση των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα κάνουν όσους έχουν ακόμα επιφυλάξεις να τις άρουν και θα καταφέρουν να ταράξουν τα νερά, έτσι ώστε να έχουμε επιτυχία στις επιδιώξεις μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε βελτιώσουμε το έργο μας εντός του Eurogroup και έτσι ώστε ε, να ε, υιοθετήσουμε ε, αυτά τα οποία επιθυμούμε. Να βάλουμε τη διάσταση της επιθυμίας δηλαδή στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε και υλοποιούμε. Έτσι ώστε να ολοκληρωθεί πραγματικά το ενιαίο νόμισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλύψατε όλα τα θέματα. Αγγίξατε όμως ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. στο οποίο υποχρεούμε τώρα να σας απευθύνω παρατήρηση και ερώτηση. Την ιδιαίτερη υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωζώνη καλύτερα, που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο της σε σχέση με ορισμένους ηγέτες κρατών, δεν θέλω να δώσω ονόματα, αλλά και σε σχέση με την κρίση που προξενούν άκρες ε, εθνικιστικές, λαϊκιστικές ε, τοποθετήσεις. Ενώ ταυτόχρονα πολιτικές κρίσεις σε ορισμένες χώρες καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Πολλά είναι τα θέματα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Ξαναδίνω το λόγο στον Πρόεδρο κύριο Γκουαλτιέρη για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ να λαμβάνω πρώτα να μιλήσω ως ομιλητής, να κάνω την παρέμβασή μου. Εάν λοιπόν συζητούμε το τι μένει ακόμα να γίνει για να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, στην παρούσα 20η επέτειο, 20 ίσως θα είναι σκόπιμο να κοιτάξουμε και πώς βλέπουμε το ευρώ, πώς κρίνουμε την επιτυχία του, εγώ τουλάχιστον, εμείς τουλάχιστον φαντάζομαι, και όλα τα επιτεύγματα που έχει φέρει, όλα τα κέρδη που έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Και αυτό νομίζω γιατί ε, πρέπει καταρχάς να εξεταστεί το ευρώ ως ένα ισχυρό οικονομικό εργαλείο, αλλά όχι μόνο ως οικονομικό, αλλά ως ένα εγχείρημα πολιτικό όσο και οικονομικό. Έτσι λοιπόν το ευρώ είναι ένα απαραίτητο συμπλήρωμα της εσωτερικής αγοράς. Έχει συμβάλει στην εξαιρετική ανάπτυξη του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου, άμεσα ή έμεσα, διότι πρέπει να θυμάμαστε ότι ένα μοντέλο που θα στηριζόταν σε, μια, σε ένα συγκριτικό ανταγωνισμό αναμφισβήτητα και αναπόφευκτα θα οδηγούσε σε ένταση ε, και ανάδειξη νέων ανταγωνισμών μεταξύ των κρατών μελών που άρα θα εμπόδιζε την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Άρα βλέπουμε ότι το ευρώ έχει εξασφαλίσει άνευ προηγουμένου ε, ολοκλήρωση ή ενοποίηση των αλυσίδων ε, αξίας που ήταν και κινητήρα για την ιστορική ε, αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγική, τον παραγωγικό κλάδο της Ευρώπης. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε και την άλλη διάσταση, την διάσταση της οικονομικής πολιτικής, την πολιτική σημασία του ευρώ. Ένα νέο νόμισμα λοιπόν και πιστεύω ότι οφείλουμε να το πούμε αυτό σε μια τέτοια συζήτηση για το τι σημαίνει εθνικό νόμισμα και τι δεν είναι εθνικό νόμισμα. Ένα νέο νόμισμα λοιπόν πρέπει να εξεταστεί ως προϋπόθεση για τη διαφύλαξη και την ανάκτηση της νομισματικής επιμερισμένης κυριαρχίας. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τις εξωτερικές πιέσεις, γιατί είναι προφανές ότι μετά την κρίση του συστήματος ε, της τάξης του Bretton Woods και της παγκοσμιοποίησης μόνο ένα ενιαίο νόμισμα θα μπορούσε να διαδραματίσει με επάρκεια το ρόλο ενός παγκοσμίου απήχηση νομίσματος και να στηρίξει τις εθνικές οικονομίες παρότι πολλά ακόμα έχουν να γίνουν όπω είπε ο κ. Μοσκοβησίος προ το διεθνή ρόλο του ευρώ και εσωτερικά το ευρώ έχει επιτρέψει σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη να έρθουν σε ανταγωνιστική ισότιμη, ανταγωνιστικά ισότιμη βάση σε σχέση με την οικονομική του και νομισματική πολιτική χωρίς το ευρώ τα περισσότερα κράτη-μέλη και κυρίω τα πιο ευάλωτα μεταξύ αυτών δεν θα ήταν περισσότερο αλλά λιγότερο, δεν θα είχαν περισσότερη, αλλά λιγότερη νομισματική και οικονομική κυριαρχία και θα ήταν αναγκασμένα να ακολουθούν ακολουθούν τις νομισματικές επιλογές των μεγάλων, της, ε, των μεγάλων νομισμάτων. Έτσι λοιπόν το ευρώ μπόρεσε να αποτελέσει ταυτόχρονα και μια θεμελιώδη προϋπόθεση για την προστασία και την επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού και οικονομικού μοντέλου σε μια μεταλλασσόμενη περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και πολιτικό ορόσημο για μια ε, ε, πολιτική πολιτικό ακρογωνιαίο λίθο και μια ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση. Ταυτόχρονα όμως αυτή η οικονομική κρίση που έχουμε περάσει έχει δείξει και τις αδυναμίες του οικοδομήματος της ε, ΟΝΕ, ε, δηλαδή ότι αν δεν υπάρχουν επαρκή ε, ρυθμιστικά πλαίσια κινδυνεύουμε από κατακαιρματισμό, ε, ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα ενιαίο δημοσιονομικό για τις εγγυήσεις, ε, η ρευστότητα. Είδαμε τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν όταν δεν είμαστε σε θέση εγκαίρως να δώσουμε με μηχανισμούς σταθεροποίησης απάντηση στην κρίση. Είδαμε μείγματα πολιτικής που είχαν περισσότερο στόχο την εξυγένση του προπολογισμού και που ως εκ τούτου οδήγησαν σε μια δεύτερη φάση της ύφεση. Έτσι λοιπόν η Νομισματική Ένωση είναι ανεπαρκής, είναι ατελής ακόμη. Ναι, υπήρξαν κάποιες εσφαλμένες αποφάσεις επίσης αλλά έχει δείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα το ευρώ και αυτό χάρη και στην πολιτική βούληση για τη διαφύλαξη της ε, ακεραιότητάς του αλλά και της ευελιξίας με ένα κοινό λοιπόν εργαλείο διαχείρισης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μπόρεσε να αξιοποιήσει πλήρως τις προνομίες της ε, δεσμευόμενη να κάνει ό,τι χρειαστεί για την προστασία της ακεραιότητας της Ευρωζώνης με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα που αποδεικνύει ότι και με κόστος μηδενικό ευρώ Έχουμε εξαιρετική απόδοση σε μέτρα όπως αυτά της πρότασης της Ντοβίλ αντί για τα ε, συστήματα τα οποία θα καθυστερούσαν ακόμα περισσότερο. Έχουμε λοιπόν ένα μηχανισμό για την εξυγίανση, έχουμε την ποσοτική χαλάρωση, η οποία ήταν θεμελιώδης για να αποφευθεί ο πληθωρισμός και να διευκολυνθούν οικονομικές ε, συνθήκες σε όλη την Ευρωζώνη. Βελτιώσεις που τώρα μας δίνουν καλύτερα οικονομικά στοιχεία, μια ευρεία και στεναρή οικονομική ανάκαμψη και έστω και αν τώρα η οικονομία επιβραδύνεται, έχουμε τα θεμελιώδη στοιχεία στη διάθεσή μας με κάποια ενδεχομένω επεκτατική δημοσιονομική τάση που ίσως να μην είχε προβλεφθεί αλλά πάντως υφίσταται και πολύ καλά υφίσταται και ξεπερνάει η δημοσιονομική ενίσχυση στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ε, ωστόσο, αν δούμε τη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε, τότε προφανώς είμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου και χρειάζεται να κάνουμε αποφασιστικά βήματα για να ολοκληρωθεί ο ναι, ιδιαίτερος ε, σε σχέση με την κρίση στο δημόσιο χρέος στις ανισότητες, στην ε, ανεπαρκή ανάπτυξη παραγωγικότητας, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλές επενδύσεις, συνεχιζόμενες κοινωνικές αδικίες και ανισότητες, ε, ζητήματα ανθεκτικότητας σε ενδεχόμενη νέα κρίση. Βλέπουμε και χαίρομαι που όλοι στέλνουμε το ίδιο μήνυμα ότι κανείς δεν επαναπάβεται και όλοι επαγρυπνούμε και λέμε ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πού πρέπει να αναλάβουμε δράση. Συμμερίζομαι και εγώ τι προτεραιότητε που έχουν ε, περιγραφεί, αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω κάποια στιγμή από αυτά του κύριου Σαντέρου. Έχουμε λοιπόν βεβαίω την ανάγκη να ολοκληρώσουμε την ΟΝΕ μαζί με την κεφαλαιακή αγορά. Θα είναι σαφέ νομίζω συν το χρόνο πόσο σημαντικό είναι αυτό και για την ανάπτυξη, τη σύγκληση, την ανθεκτικότητα τη οικονομία Χρειάζεται να επιταχύνουμε το πακέτο για το περιορισμό του κινδύνου. Έχουμε συμφωνία για το backstop. Ε, Βεβαίω πρέπει αυτό το backstop, ο εναλλακτικό μηχανισμό δηλαδή, να είναι εναλλακτικό μηχανισμό και όχι μνημόνιο. Αλλά πρέπει να δώσουμε τώρα απαντήσει και για, το τρίτο, για τον τρίτο πυλώνα, για το σύστημα το ασφαλιστικό διασφάλιση. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να περιορίσουμε τους κινδύνους σε σχέση με τη χρήση κεφαλαίων και ρευστότητα στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, κάτι που είναι απαραίτητο για μια τραπεζική ένωση. Η ομάδα υψηλού επίπεδου θα κάνει τη δουλειά τη, περιμένουμε να τη δούμε. Θα συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ε, ω προ ε, το κίνδυνο, τον περιορισμό του κινδύνου και τι απαιτήσει περιορισμού του κινδύνου, κρατικό χρέο δηλαδή και άλλα, που ίσω αν είμαστε υπερβολικοί στι απαιτήσει μα μπορεί να οδηγήσει περισσότερο σε αύξηση του κινδύνου παρά σε περιορισμό του κινδύνου. Εργαλεία διαχείριση κινδύνου, ο μηχανισμό κάνεις πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν οι προληπτικές γραμμέ, γραμμές, δημοσιονομικές γραμμές. Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν οι προνομίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά πρέπει να είναι ο ESM ε αυτόνομος και στη συνέχεια φτάμε στην ανάγκη για ένα ειδικό εργαλείο δημοσιονομικό για την Ευρωζώνη, γιατί όταν έχουμε κοινό νομίσμα, οπωσδήποτε έχουμε και ιδιάζουσες ανάγκες, τι οποίε θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε με ένα ιδιάζον ιδιαίτερο εργαλείο δημοσιονομικό. Χαίρομαι που πια έχει μπει αυτή η δουλειά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τη Ευρωζώνη. Επιτρέψτε όμω πολύ σύντομα να δώσω απάντηση στο μέλο Αντένου λέγοντα τα εξή. Παρατηρήσει πολύ σημαντικέ εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξεκινώ λέγοντα ότι ναι, συμφωνούμε πω αυτό το ειδικό δημοσιονομικό εργαλείο πρέπει να εγγράφεται μέσα στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και άρα να υπάγεται στην κοινή δημοσιονομική διαδικασία. Δεύτερον, και είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με συμπληρωματικέ λειτουργίε, λειτουργίε, οι οποίε δεν μπορούν να ε, βγαίνουν από την, συνή... από την κοινή πολιτική για τη σύγκληση, για την ε, συνοχή. Ε, πρέπει να διατηρηθεί δηλαδή αυτή η ισορροπία μεταξύ περιφερειών της Ευρωζώνης ή περιφερειών εκτός Ευρωζώνης. Επομένως επιπλέον χρήματα θα χρειαστούν και όχι επανανάπτυξη, επαναχρήση φυσταμένων κονδυλίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και τρίτον, χρειάζονται και οι δύο λειτουργίες. Και οι δύο λειτουργίες και η σύγκληση είναι πολύ ωραία, αλλά και η σταθεροποιητική λειτουργία, η οποία έχει κέρια σημασία εάν κοιτάξουμε τα διδάγματα της κρίσης. Η δημοσιονομική ε, υποστήριξη μπορεί να συνδυαστεί με ένα είδος ε, ισοστάθμισης με την σταθεροποίηση. Αλλά δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι η σταθεροποιητική λειτουργία έχει τεράστια σημασία για τη λειτουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης και μόνο η σύγκληση στην οικονομική πολιτική δεν μπορεί να αρκεί. Και επίσης, αν μου επιτρέπει ο χρόνος, θα ήθελα να συμπληρώσω στο, σε αυτά που είπε και ο Πιέρ Μοσκοβισή, ότι δεν είναι δυνατόν το ευρώ και το μέλλον του να, κληθεί, να κρυθεί στο ύψος του προϋπολογισμού. Πρέπει να υπάρχουν τα εργαλεία αυτά και ταυτόχρονα πρέπει να μας απασχολήσει και η βελτίωση του δημοσιονομικού πλαισίου. Χτες συζητήσαμε επί μακρόν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, ε, πώς μπορούμε να έχουμε πιο απλά δημοσιονομικά πλαίσια, πώς μπορούμε να έχουμε λιγότερο εκτεθειμένα στους κυκλικούς κλειδονισμούς συστήματα και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα με ένα ειδικό εργαλείο δημοσιονομικό της Ευρωζώνης που οπωσδήποτε πρέπει να προχωρήσει. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλησίου και για τη δημοκρατική διάσταση τελευταία παρατήρηση απολύτως ουσιώδη και χαίρομαι για τα όσα είπε ο Πιέρ εδώ. Έχουμε μια χρυσή αρχή, χρυσή αρχή που μπορεί να μας διαφωτίσει και εσάς και εμάς. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ε, στεναρή δημοσιονομικό στεναρός δημοσιονομικός έλεγχος στα δημοσιονομικά της Ευρωζώνης πρώτον και απαραίτητον και δεύτερον κάθε απόφαση θα πρέπει να εκτίθεται στον απαραίτητο βαθμό της κοινοβουλευτικής επίβλεψης ή του ελέγχου ανάλογα με το επίπεδο της ε, διακυβέρνησης, της διαχείρισης. Επομένως, αν πρόκειται για κονδύλια εθνικά, έλεγχος από το Εθνικό Κοινοβούλιο, αν πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια, έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδάλλως θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το δημοκρατικό ε, χάσμα που έχουμε και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στον πολίτη γιατί χρειαζόμαστε και άλλα κονδύλια. Πρόκειται για έναν πιθανός αγαθό κύκλο αλλά πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά στους φίλους του Συμβουλίου. Μερικές φορές μας περιγράφουν σαν αντίπαλα στρατόπεδα, σαν να ε, διεκδικούμε εμεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια αρμοδιότητες. Όχι, τουναντίον, αντίον, στο, από την ίδια πλευρά αγωνιζόμαστε. Θέλουμε ένα δημοκρατικό έλεγχο, ένα σύστημα νομοποίησης και δημοκρατικής λογοδοσίας σε εθνικό όπω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν συνεχίσουμε το διάλογο αυτό, μπορούμε, πιστεύω, ενωμένοι να πιέσουμε για μια δημοκρατική διάσταση αυτού του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο πάλι στον κύριο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη, ο οποίος θα συντονίσει την ε, σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ, λέει ο Σκουαλτιέρη. Γκουαλτιέρη. Γνωρίζετε τους κανόνες, να μην τους ε, επαναλάβω. 12 και 42 μου είπαν ότι πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει, γιατί θα έρθει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριο Ντομίγκος, Πορτογαλία, ΕΛΚ, είναι ο πρώτος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εδώ βρίσκομαι. Είμαι από το PSD. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ευχαριστώ πολύ. 20 χρόνια του ευρώ. Υπάρχουν λόγοι για ικανοποίηση. Πολλοί βουλευτές, ευρωβουλευτές ε, είχαν στοιχηματίσει ότι δεν θα επιζούσε το ευρώ και όμως επέζησε. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν για να έχει μεγαλύτερη αντοχή σε κρίση στο ευρώ. Μετά από τα τελευταία γεγονότα, την κρίση, οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν θέλησαν να αλλάξουν πολύ τα πράγματα. Το είπαμε και σήμερα. Σημαντικά μέτρα. Όμως, προσοχή. Συγχρόνως, στον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης έχουμε ελάχιστη πρόοδο. Πρόκειται για την εγγύηση καταθέσεων. Είναι σαν να χτίζουμε ένα σπίτι χωρίς να έχουμε έναν βασικό τοίχο, ένα φέροντα τοίχο. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, στην ε, διάσκεψη κορυφής, απογοητευτήκαμε, γιατί τίποτα δεν έγινε για να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μιλήσαμε για ανισότητε, μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα από το να έχει διαφορετική αξία το ευρώ σε κάθε χώρα, το να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασία για να λυθεί αυτό το πρόβλημα του μηχανισμού εγγυήσεων καταθέσεων, είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα λύσει το πρόβλημά μας. Απλώς είναι μια διέξοδος ε, προς τα μπρος. Αποφεύγουμε αυτό που πραγματικά χρειάζεται, μια πραγματική μεταρρύθμιση. Αφήνουμε ένα σπίτι χωρίς να έχει τελειώσει. Και η επόμενη κρίση θα έρθει κάποια στιγμή. Ο κύριος Βότσης από την Κύπρο, παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, το ευρώ επιβίωσε της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του. Εν τούτης, η χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε τις θεμελιώδεις και εγγενείς αδυναμίες του. Σε πολιτικό επίπεδο σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος για τη διόρθωση των αδυναμιών του ευρώ. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η οικονομική κρίση ενέτεινε περαιτέρω τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ του πλούσιου βορρά και του χρεοκοπημένου νότου. Η έλλειψη αναδιανομής του πλούτου και επιμερισμού των βαρών εν καιρό κρίσης κατέδειξε την έλλειψη έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. Το χάσμα του κατακεφαλήνα ΕΠ και των ρυθμών ανάπτυξη τη οικονομία τη χώρα τη Ευρωζώνη οξύθηκε περαιτέρω. Οι 19 χώρε μέλη τη Ευρωζώνη εξακολουθούν να μην έχουν στη διάθεσή του επαρκή εργαλεία για επίτευξη τη οικονομική σύγκληση και για προσέλκυση επενδύσεων. Τώρα που βελτιώθηκαν οι κοινωνικο-οικονομικέ συνθήκε, όχι μόνο δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, αλλά πρέπει να αξιοποιήσουμε το momentum για επιτάχυση της υλοποίησης των απαραίτητων θεσμικών μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκληση, να διορθωθούν τα ευάλωτα σημεία και να εδραιωθούν οι συνθήκε βιώσιμη ανάπτυξη, προόδου και κοινωνική ευημερία. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να δώσουμε κίνητρα στι χώρες που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για όλες τις χώρες. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ολοκλήρωση της ΩΝΕ, είπαμε όλοι και θα ακούσετε και στη συνέχεια για τον περίφημο μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων που πρέπει να προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις, η ολοκλήρωση λοιπόν τη Τραπεζική Ένωση, τη ενιαία αγορά και τη Ένωση Κεφαλαίου Αγορών είναι απαραίτητε προποθέσει για την ενίσχυση του διεθνού ρόλου του ευρώ. Τέλο, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα αποτελέσματα τη έρευνα που έχει αναφέρει ο Επίτροπο Μοσκοβισή, που λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν μετά τα 20 χρόνια επιτυχημένο το εγχείρημα ευρώ. Βεβαιότητα όμω μπορούμε ακόμα καλύτερα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαδημούλης, Ευρωβουλευτής Γκουε. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχοντας 20 χρόνια ευρώ θα πρέπει να δούμε όχι μόνο τι έχει επιτευχθεί, αλλά κυρίως τι λείπει και τι πρέπει να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Γιατί οι αριθμοί δείχνουν από τη μια ανθεκτικότητα του ευρώ, αλλά από την άλλη και κατασκευαστικά λάθη, τα οποία έχουν οδηγήσει στην αύξηση των ανισοτήτων και των κοινωνικών και των περιφερειακών. Και επειδή η αύξηση των ανισοτήτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρέφει την ακροδεξιά και υπονομεύει την μακροημέρευση του ευρώ και επειδή δεν μπορεί να σταθεί ένα κοινό νόμισμα χωρίς μια κοινή πολιτική ενοποίηση και δημοκρατική λογοδοσία και περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη συνοχή, θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα. Κύριε Σεντένο, η διεθνής διαφάνεια με την πρόσφατη έκθεσή της ζητάει από το Eurogroup περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη δημοκρατική λογοδοσία. Δεν μπορούν τόσο σοβαρά θέματα να αποφασίζονται πίσω από κλειστές πόρτες. Είσαστε υπέρ του να λογοδοτείτε όχι μόνο στα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, σημερίζομαι, κύριε Μοσκοβισή πολλές από τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας. Αλλά μπορείτε να μου πείτε γιατί μερικές δεκάδες δημοσιογράφοι, whistleblowers, ανακαλύπτουν μεγάλα σκάνδαλα φοροδιαφυγής και δεν μπορούν αυτά να τα ανακαλύψουν και να επιβάλλουν ποινές οι υπάρχοντες ευρωπαϊκοί θεσμοί. Γιατί τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που χάνονται από τους κρατικούς και από τον κοινοτικό προϋπολογισμό από τη φοροδιαφυγή των πλουσίων και των μεγάλων πολυεθνικών τα πληρώνουν με υπερφερολόγηση οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν απαντήσεις γιατί έχουμε μια ατελή οικονομική ένωση, ατελή νομισματική ένωση, ατελή τραπεζική ένωση και πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα μπρος. Thank ευχαριστώ. Φόρτι Ιταλία, e Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εορτάζουμε την 20η ε, επέτειο από την εισαγωγή του ευρώ. Οι πανηγυρισμοί αυτοί οφείλονται στο ότι ύστερα από 25 η απο την εισαγωγη του ευρω υπάρχει ακόμα το ευρώ. Ναι, μπράβο. Υπάρχει ακόμα το ευρώ, όντω. Επιτυχία όμω. Ήταν επιτυχία για όλου. Θα έπρεπε να έχει χαρακτηριστεί από σύγκληση και συνοχή. Κι όμως αντιθέτως βλέπουμε απόκληση και διχασμούς μπορούμε να δούμε πολύ εύκολα ένα στιγμιότυπο των αποκλήσεων αυτών. Οι οικονομικές επιδόσεις μετά την κρίση, οι οικονομικές επιδόσεις της Ευρωζώνης είναι χειρότερες από τις υπόλοιπε ανεπτυγμένε οικονομίες. Ακόμη και τώρα που μιλάμε. Χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν εισαγάγει το ευρώ έχουν υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξη από τι χώρε τη Ευρωζώνης. Ήταν επιτυχή η εισαγωγή του ευρώ για την Ελλάδα. Ήταν επιτυχία για την Ιρλανδία. Ήταν επιτυχία για τη Γαλλία. Για να δούμε, η Ιταλία τι είδε. Άξιζε πράγματι να κάνουμε και πανηγυρισμούς σε 20 χρόνια. Ανάπτυξη 0. 3% έστω, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μηδενική. Έχει την υψηλότερη ανεργία στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας δεν υπάρχουν ασφαλή ε, στοιχεία ενεργητικού για, τις, ε, για, την, ε, για τους καταθέτες. Έχουν επιβληθεί κανόνες μετά την διαφορετική ρύθμιση και διάσωση των τραπεζών στις περιόδους της κρίσης. Υψηλότερο κόστος δανεισμού, 3% στην Ιταλία σχέση με τη Γερμανία. Τι μιλάμε λοιπόν για νέο νόμισμα όταν υπάρχουν τόσο σημαντικές αποκλήσεις σε κόστος δανεισμού. Ε, σταμάτησαν να αυξάνονται οι μισθοί, οι πραγματικοί μισθοί και μειώνονται κιόλα. Και το πληρώνουμε αυτή την επιτυχία, την πληρώνουμε ακόμα. Και όχι μόνο η Ιταλία. Οι προσεχεί εκλογέ, λοιπόν, νομίζω θα επιτρέψουν τον πολίτη να αποστείλει το μήνυμα τη ευτυχία που αισθάνεται και στη Γαλλία και στη Γερμανία ακόμα για την διαχείριση τη Ευρωζώνη. Μιλάτε συχνά για λαϊκισμό, του λαϊκιστές, ω εχθρού σαν να είναι μόλυνση, ρήπανση σε έναν υπέροχο κόσμο. Και στις εγωγικές σας παρατηρήσεις, α, πρέπει να καταπολεμήσουμε την ανάδειξη των λαϊκιστών. Όμως δεν είναι αυτό. Ο λαϊκισμός είναι μια δημοκρατική αντίδραση των ευρωπαϊκών λαών, των ευρωπαίων πολιτών, έναντι μια ελίτ που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Πιστεύω λοιπόν οι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων που θα έρθουν στο μέλλον σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο και αυτοί που θα έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τι προσεχέ εκλογέ. Θα είναι άλλοι, θα το κάνουν καλύτερο το Κοινοβούλιο, θα το κάνουν διαφορετικό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε. Το οικονομικό κόστο θέλαμε να είναι χαμηλότερο. Ο κύριο Βαλούρα, Ελλάδα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Την πρωτοχρονιά του 1999 που εισήχθη το ευρώ, πολιτικοί και αναλυτές έκαναν λόγο για μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις του 20ου αιώνα. Όποιος τότε μίλαγε για τα δομικά προβλήματα που μπορεί να είχε εισαγωγή του ευρώ, με τον τρόπο που έγινε θεωρώνταν κασάδρα, ακόμα κι αν ήταν νομπελίστας οικονομικής επιστήμης. Σήμερα θυμίζω του στόχου τη Ενωσματική Ένωση. Πρώτον, ταχύτερη σύγκληση των οικονομιών τη Ευρώπη και δεύτερον, βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. 20 χρόνια μετά από τη μεγάλη οικονομική κρίση της Ευρωζώνης, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει σε κάποια σημεία όπως τη διευκόλυνση των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών, τις διακρατικές ροές κεφαλαίων και κάνοντας το ευρώ βάση για μια πιο οικονομικά ισχυρή και με κοινωνική και περιφερειακή συνοχή Ευρώπη. Όμως, κατά τη διάρκεια της, δεκα... της χρυσής δεκαετίας του ε, ευρώ, που κανείς δεν μπορούσε, δεν τολμούσε να αφισβητήσει το νέο νόμισμα, είναι χαρακτηριστικότατο το 1999 έως το 2008 οι διακρατικές απαιτήσεις των τραπεζών της Ευρωζώνης σε 10, από 1-3 σε 13 ευρώ με αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων τον υπερδιπλασιασμό του διευρωπαϊκού εμπορίου. Όμως, κύριε Πρόεδρε, με την οικονομική κρίση διαφάνηκαν οι δομικές αδυναμίες της Νομιαντικής Ένωσης και του ευρώ και, δεν, και συνειδητοποιήσαμε τότε ότι οι βασικοί στόχοι της ΟΝΕ όπως η σύγκληση, η συνοχή, η ανάπτυξη είχαν ξεχαστεί ή επαόριστον αναβληθεί ταυτόχρονα οι μηχανισμοί πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων είτε δεν υπήρξαν είτε δεν λειτουργήσαν. Για μια χώρα, για μια χώρα σαν την Ελλάδα θυμίζω ότι ακόμα και πρόβλημα εισαγωγής της στη ζώνη του ευρώ υπήρξε και ισοτιμία αλλά είναι μια άλλη συζήτηση θα την κάνουμε άλλη φορά. Το θέμα είναι όμως κύριε Πρόεδρε ότι αν μάθαμε και πρέπει να μάθουμε ότι εάν θέλουμε βάθηση του, του, του, της ΟΝΕ θα πρέπει να μιλήσουμε και το δημοκρατικό έλεγχο και τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν μπορεί ένα όργανο σαν το Eurogroup το οποίο παίρνει σημαντικό τις αποφάσεις για τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων να μην έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και πολλές φορές τεχνοκράτες να μιλάνε και να κανονίζουν την πολιτική των λαών της Ευρώπης. Υπάρχουν λοιπόν δομικά προβλήματα και τελειώνοντα κύριε Πρόεδρε λέω ότι σκληρέ, πέραν των δομικών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, των σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών με, μαζί με τις δομικές, αλλά, ε, ε, ε, ε αύξησαν τα επίπεδα φτώχειας και ανεργίας τα τελευταία χρόνια τροφοδοτώντας ακροδεξιές και αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερνάντες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Σεντένο, τον πρόεδρο του Eurogroup. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει προτάσεις για την ενίσχυση της συνοχής και της σύγκλησης στην Ευρωζώνη. Ε, η Ευρωμάδα δεν έκανε καμία πρόταση Κύριε Πρόεδρε, λέτε ότι τον Ιούνιο θα υπάρξει μια πρόταση. Οι εκλογές προβλέπονται 26 Μαΐου, οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα τον Ιούνιο και ίσως γι' αυτό δεν ήσασταν στο Στρασβούργο στη συζήτηση όταν συζητήσαμε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του ευρώ. Αλλά τουλάχιστον απαντήστε μου εδώ σε μια ερώτηση κύριε Σεντένο για το καλό του προπολογισμού του ευρώ, ο μηχανισμός σταθερότητας επενδύσεων είναι κάτι το οποίο σας βρίσκει σύμφωνο. Συμφωνεί το Eurogroup με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τα 30 εκατομμύρια για το μηχανισμό αυτό, πρικοδότηση. Πώς βλέπετε εσείς την χρηματοδότηση, με τι πόρους. Δέχεστε, συμφωνείτε ότι τα κέρδη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ήδη πόροι και ως εμβριακή μορφή ενός προπολογισμού της Ευρωζώνης. Ελπίζω ότι μπορείτε, αν μη τι άλλο, να μου απαντήσετε απλά και ξεκάθαρα σήμερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μάλσκα Βίνκαμαν, Γερμανία, EFDD. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η επίκρισή μου είναι ότι με ωραία λόγια φαίνεται να εξαίρεται η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, ενώ ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας διαπιστώνει έλλειμμα 25 δισεκατομμύρια για τον εθνικό προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι επιτυχημένη η εισαγωγή του ευρώ, η λειτουργία του ευρώ, όταν έχουμε δουλέψει με αρνητικά επιτόκια χρόνια, όταν ο μικροκαταθέτης έχει χάσει την αξία ε, του χρήματός του. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι ο μέσος πολίτης έχει δει μάλλον αρνητικές συνέπειες με τα αρνητικά επιτόκια που τον οδηγούν και σε προχωρημένη ηλικία πολύ συχνά στη φτώχεια, άρα κάτι το μη αναστρέψιμο. Και γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωζώνη ήταν ε, ε, επιζήμια για τον μέσο πολίτη. Πολλά είναι τα κράτη που είχαν πρόσβαση σε, πολύ φθηνά, σε πολύ φθηνές πιστώσεις όπως η Ιταλία με 100 δισεκατομμύρια που δεν μπορεί να αποπληρώσει, με εκατοντάδες δισεκατομμύρια που δεν μπορεί να αποπληρώσει και έτσι επιβαρύνει τώρα το σύστημα λόγω των, ε, της υπερβολικής χρέωσης και έκθεσης των ε, τραπεζών της Ιταλίας και που καλείται μετά η Γερμανία να διασώσει ε, μάλιστα με μια πρόταση η οποία οδηγεί από, μονο, από ομοφωνία των Συμβούλων να λαμβάνει αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Δηλαδή ακόμα περισσότερο τίθεται σε κίνδυνο η κατάθεση του Γερμανού μικροκαταθέτη. Και για να ολοκληρώσω, ε, το να μιλάτε για λαϊκισμούς και ακροδεξιά όταν απλώς τυπώνετε μία άποψη διαφορετική σημαίνει και αδυναμία αποδοχής της δημοκρατικής αντιπαράθεσης. Όταν δεν το κάνετε αυτό, όταν δεν το κάνετε αυτό αποδεικνύεται ε, ότι απλώς έχετε χάσει κάθε έννοια ευγένειας δημοκρατικού διαλόγου το να περιγράφετε δηλαδή τον αντίπαλό σας τον πολιτικό ως λαϊκιστή και ακροδεξιό ο κύριος Γουαλτιέρη. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται εγώ να κάνω καταδίκες ή καταγγελίες για το τραπεζικό σύστημα άλλης χώρας. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, θα πρόσεχα πολύ λοιπόν. Ωστόσο τώρα έχουμε το εξή ζήτημα, έχουμε περιορισμένο χρόνο, ζητούν όμως και άλλοι συναδελφοί το λόγο. Επομένως μόνο εάν περιορίσουμε στο 1-1-30 λεπτά το χρόνο των παρεμβάσεων. Μπορώ να αφήσω τον κατάλογο των αγορητών. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο στου περισσότερου ε, συναδέλφου των δυνατών, αλλά πρέπει να δείξουμε ο καθένα αυτοπιθαρχία. Εάν δεν το πράξουμε, οι τελευταίοι θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Ε, Α κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να διευκολύνουμε όλου του συναδέλφου να μιλήσουν. Ο κύριο Σίλβα Περίρα, SND, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Κολτιέρη. 20 χρόνια ευρώ Άρα πρέπει να καθίσουμε και να προβληματιστούμε για το μέλλον του ευρώ και πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα επόμενες κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ποια είναι ο πορείας για το ευρώ και τι πρέπει να κάνουμε. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί μετά από τόσα χρόνια έχουν γίνει βήματα σημαντικά, δεν λέω, αλλά παρόλα αυτά όχι αρκετά, παραμένουν πάρα πολλά να γίνουν. Το θέμα έχει να κάνει ακριβώς με το αδιέξοδο που έχουμε μπροστά μας. Το πώς δηλαδή θα κατανέμουμε τους κινδύνους. Κάποιοι είπαν ότι αντίθετα από αυτό που λέει ο κύριος Φερνάντες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν αντιστάσεις για να, δώσουμε, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω για τη μεταρρύθμιση του ευρώ. Ότι υπάρχει δηλαδή μία ατζέντα για μείωση του κινδύνου που δεν προχωράει, που δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Αυτό το αδιέξοδο πρέπει να το ξεπεράσουμε. Έχοντας μειώσει το χρέος και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τώρα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση του ευρώ. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να κατανείμουμε τους κινδύνους. Κροατία, Έλκα, Πέρσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ τα 27 χρόνια που έχουμε το ευρώ. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Η Κροατία, που είναι το τελευταίο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει βάλει μπροστά μια στρατηγική για να ενταχθεί στο ευρώ. Και είναι αλήθεια ότι χρειάστηκε να κάνουμε πολλά. Οι απαιτήσει ήταν πολλές. Το 2016 ήταν και η πρώτη χρονιά όπου μπορούσαμε να πούμε ότι ολοκληρώσαμε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να ε, συμμετέχουμε κι εμείς στον ε, μηχανισμό σε δεύτερο στάδιο. Το έλλειμμα είναι κάτω από το 3% του ΕΠ και το δημόσιο χρέος επίσης μειώθηκε πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε, με πιο γρήγορο ρυθμό. Συνεπώς, τα δημοσιονομικά μας είναι σταθερά. Αυτό το οποίο μας διακρίνει από άλλους και μας δίνει πλεονέκτημα είναι το ότι... Ε, πέντε δευτερόλεπτα έχετε ακόμα διακόπτει ο Πρόεδρος. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο οι υπόλοιποι. Αλτό. Ε, Φιλανδία, πράσινη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο στην ευθύνη που έχει κάθε χώρα μέλος για τις μεταρρυθμίσεις στον προπολογισμό της. Ε, πολλές χώρες, ε, ο ιδιωτικός ο τομέας βρίσκεται σε μεγάλη χρέωση. Οπότε είναι ευθύνη αλλά και προνόμιο των χωρών μελών. Και αυτό μας οδηγεί να προβληματιστούμε και για το δίδυμο έλλειμμα και πλεόνασμα. Είμαστε σε ένα διέξοδο. Πρέπει να τηρούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες στις χώρες μέλη βλέπουμε ότι υπάρχουν σαφείς ορισμοί και κανόνες. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, σταθεροποίησης που να είναι αποτελεσματικός. Αλλιώς έχουμε κανόνες οι οποίοι δεν τηρούνται και οι οποίοι συνεχώς παραβιάζονται, κάτι το οποίο είναι αρνητικό για όλους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μαργκερίτα Μάρκες, Πορτογαλία. Σοσιαλιστές, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω ευχαριστώντας πρώτα απ' όλα όλους για τις παρεμβάσεις. Ε, κύριε Σεντένο, ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο με τον οποίο επιμένετε ε, για τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου και μιλάτε για τις ευθύνες και πώς στην πράξη θα υλοποιήσουμε τον χάρτη πορείας που, στον οποίο κατέληξε η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου. Τώρα, ένα πράγμα τονίστηκε και αυτό είναι ότι οι χώρες χάνουν την ικανότητά τους υποτίμησης των νομισμάτων τους μεν, από την άλλη μεριά έχουν διαφορετική πρόσβαση όσον αφορά τα επιτόκια και άρα έχουν διαφορετική πρόσβαση στις αγορές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν δημιουργηθούν ειδικοί μηχανισμοί, τότε οι προϋποθέσεις που δημιούργησε το ευρώ οδηγούσαν σε απόκληση και όχι σε σύγκληση. Όλοι καταλαβαίνουμε πως η κρίση του 2007 και 2008 είχε σαν ε, συμπέρασμα το ότι αν δεν είχαμε το ευρώ η κρίση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, πολύ χειρότερη. Γι' αυτό θέλω να αντιδράσω σε αυτά που είπε κάποιος από τη Λίγκα που πήρε το λόγο πριν από μένα και αναφέρθηκε στο ευρώ. Σίγουρα και ανεξάρτητα από το ότι είναι βάλωτο ε, το ευρώ είναι επιτυχία. Σήμερα αντιμετωπίζει δύο τεράστιες προκλήσεις. Πρώτον, να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ και όλοι οι πυλώνες και το υπενθύμησε ο κύριος Μοσκοβισή είπε για τον τρίτο πυλώνα και από την άλλη μεριά να φτιάξουμε μια δημοκρατική ΟΝΕ που να μπορεί να ελέγχει δημοκρατικά τα εθνικά κοινοβούλια δηλαδή και το Ευρωκοινοβούλιο να μπορούν να κάνουν δημοκρατικό έλεγχο. Μια Ιταλία ΕΝΕΦ. Thank you, Mr. President. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι παραδέχονται και παραπονιούνται και δέχονται το γεγονός ότι η Ευρωζώνη δεν έχει λειτουργήσει όπως θα ήταν επιθυμητό. Ο ρόλος της ως κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη ε, συνοψίζεται στα βασικά αριθμητικά στοιχεία. 1,29 ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης το 11 με 13 και στις χώρες εκτός ευρώ ήταν πάνω από 2%. Είναι λάθεια όλα αυτά ε, και ελαττώματα και δεν μας ε, είναι το αποτέλεσμα της αποπληθωριστικής μεροληψίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή υπάρχει μεροληψία με αυτή την αιμονή για χαμηλό πληθωρισμό και ε, ε, ε δεν μπορούμε να έχουμε υποτίμηση για να είμαστε ανταγωνιστικοί και δεν μπορούμε να έχουμε και πολιτικές αντιπαλότητες μεταξύ των κρατών μελών. Είναι λίγο δύσκολος αυτός ο τετραγωνισμός του κύκλου και πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, πρέπει να δεν μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε ασύμετρες απειλές με συμμετρικούς κανόνες. Να έχουμε προκυκλικές ε, πολιτικές στην ύφεση και αντικυκλικές επιλογές ε, στην ανάπτυξη. Εμείς οι λαϊκιστές είμαστε έτοιμοι να σταθούμε στο ύψος αυτών των προκλήσεων μετά τις επόμενες εκλογές και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει ο μηχανισμός σταθερότητας αλλά και η ρύθμιση του Eurogroup βάσει συνθήκων, το οποίο πρέπει να γίνει ένα όργανο με διαφάνεια, το οποίο να αποδίδει λογαριασμό, να δίνει λογαριασμό και θα είναι προτεραιότητές μας για την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Ο κύριος Μάρδας, παρακαλώ, τελευταίος ομιλητής. Mr. President, κάθε νόμισμα εξυπηρετεί δύο στόχους. Τις σταθερές ισοτιμίες και τη ρευσότητα στην αγορά από την άλλη όμως το πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιλεγεί αντιμετωπίζεται η ακόλουθη εξέλιξη. Ειδικότερα, εφόσον το διπλό έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επιδιώκεται να διορθωθεί μόνο με δημοσιονομικά μέτρα, δηλαδή με μείωση των δημοσίων δαπανών, καταστάσεις λοιπόν που οδηγούν στη μείωση της κατανάλωσης και των εισαγωγών, τότε για να αυξηθεί το ΕΠ χρειαζόμαστε αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Για να γίνει αυτό θα ήταν σκόπιμο να υιοθετηθεί το ακόλουθο. Να προβλεφθεί ένας μηχανισμός δημιουργίας ρευστότητα στην βραχυχρόνια περίοδο υπέρ της αγοράς των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αυξάνονται ιδιωτικές επενδύσεις και εξαγωγές. Αυτό ως αντιστάθμισμα των περιοριστικών πολιτικών που οδηγούν στη μείωση των δημοσίων δαπανών και της κατανάλωσης. Αν η Ένωση θέλει να τιμωρήσει σε εισαγωγικά ή εκτό εισαγωγικών. Μια κυβέρνηση γιατί εκτροχιάζει το κρατικό τη προπολογισμό δεν χρειάζεται απαραίτητα να τιμωρεί και την αγορά. Τιμωρία τη αγορά με έλλειψη ρευστότητα στη βραχυχρόνια περίοδο οδηγεί σε στασιμότητα επενδύσεων και εξαγωγών, οξύνοντα την αβεβαιότητα που εισάγει στην οικονομία. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα διευρύνει να διευρύνει λύσει προ αυτή την κατεύθυνση δύο λεπτά για απαντήσεις. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι λίγος, το καταλαβαίνω, αλλά πρώτα ο κύριος Σεντένο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, θα είμαι σύντομος. Πρώτον, κάποιοι από εσάς μίλησαν για την ομάδα εργασίας για το IDs. Ε, υπάρχουν βουλευτές και οι Υπουργοί Οικονομικών. Ποτέ πριν το θέμα του AIDS της Υγείας καταθέσεων δεν είχε βρεθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Επίσης, πρέπει να θυμηθούμε ότι οι αποφάσεις στο Συμβούλιο λαμβάνονται από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Δεν υπάρχει έλλειψη διαφάνειας εκεί. Οπότε και αυτό δεν είναι δικιά μου προσωπική γνώμη, ήμουν ξεκάθαρο σήμερα στην παρουσίασή μου, στην ομιλία μου. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο φορές τα ίδια χρήματα, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, για τις πηγές ε, από τις οποίες θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τον προπολογισμό μας. Το βασικό μου μήνυμα σήμερα είναι ότι πρέπει να δράσουμε. Και σε μια δημοκρατία αυτό σημαίνει ψηφίζουμε. Και οι εκλογές έρχονται, φτάνουν όπου να είναι, πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε. Οπότε κάνω έκκληση σε όλους να πάνε και να ψηφίσουν. Μιλήσαμε για την ευημερία. Αυτά δεν είναι θέματα που έχουν να κάνουν για χτέ ή για σήμερα ή για αύριο. Έχουμε 50 χρόνια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η διαδικασία είναι μακρά και επιτυχής. Πολλές φορές περιορίζουμε τη συζήτηση στους καθαρούς εισφορείς και τους καθαρούς αποδέκτες. Κι όμως η διάσκεψη κορυφής του Δεκεμβρίου το έδειξε σε όλους ότι όλοι κερδίζουμε. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε από αυτή τη διαδικασία και πρέπει να συνεχίσουμε. Το ευρώ είναι ε, στα καλύτερα επίπεδά του στήριξης. Είναι το αντίθετο από τις αντιλήψεις που εκφράζουν οι ευρωσκεπτικιστές. Πρέπει να βασιστούμε στις επιτυχίες μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και να παίρνουμε αποφάσεις. Ευχαριστώ. Λέω ο κύριος Γουαλτιέρη, συνθετικά παρακαλώ και εσείς. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι όντω και εγώ σύντομος. Κοιτώντας προς τα πίσω, και κοιτώντα τι έγινε τα τελευταία χρόνια με το ευρώ, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι είχαμε πολύ χαμηλό πληθωρισμό, πολύ χαμηλά επιτόκια. Συγχρόνω, η οικονομική κατάσταση των τραπεζών μας είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Έχουν περισσότερο κεφάλαιο, μεγαλύτερη αντοχή και ο μηχανισμό ε, εποπτείας επίση έχει βοηθήσει πολύ. Νομίζω αν θέλετε τη γνώμη μου, το βασικό είναι το εξή το 80% του κόσμου στην Ευρωζώνη στηρίζει το ευρώ και πιστεύουν ότι είναι ένα καλό νόμισμα και ένα καλό μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα στρεφόμενοι προς το μέλλον θα έλεγα ότι βέβαια στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάποιες δυναμίες, κάποιες τις διορθώσαμε και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση με το ΕΝΤΙΣ, τον τρίτο πυλώνα δηλαδή της Τραπεζικής Ένωσης και την ε, Κεφαλαϊκή Ένωση και είμαστε υπέρ ενός νέου ε, μηχανισμού σταθεροποίησης της δημοσιονομικής μας ικανότητας για να αποφεύγουμε τα σύμμετρα σοκ. Όλα δεν είναι τέλεια. Ευχαριστώ, αλλά και τίποτα στον κόσμο δεν τέλειο. Ο κύριος Μοσκοβισή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση δείχνει ότι όντως το ευρώ είναι αντικείμενο δημοκρατικό, είναι αντικείμενο συζήτησης. Το ελάχιστο πρέπει να το πούμε γιατί είναι και αυτονόητο. Είναι ένα νεαρό νόμισμα, ισχυρό αλλά νεαρό και άρα είναι και ισχυρό αλλά και ατελές και μπορώ να πω απερίφραστα ότι ναι, ξέρω τι προσφέρει το ευρώ, φέρνει σταθερότητα, φέρνει προστασία, ενότητα, ισχύ. Και αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους το 64% των Ευρωπαίων που χρησιμοποιούν το ευρώ το θέλουν, είναι... το αποδέχονται και γι' αυτό και κάποιες κυβερνήσεις που κάποια στιγμή μπήκαν στον πειρασμό να αποχωρήσουν τελικά έκαναν τις προσαρμογές στις πολιτικές τους για να μπορέσουν να παραμείνουν και πρέπει και εμείς να αγωνιστούμε στο ευρώ να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικό νόμισμα, πιο πιστικό νόμισμα, ο δυναμισμός, η ανάπτυξη, η δημιουργία είναι οργασίες. οι παραδείγματι, που ξέρουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε, πρέπει να είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Είπα εισαγωγικά και γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω επαναλαμβάνοντα τους τέσσερις δρόμους τους οποίους πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον του ευρώ για να ολοκληρώσουμε το νόμισμα αυτό, τραπεζική ένωση λοιπόν που πρέπει να ολοκληρωθεί και ο Λούις Δεκίντους που ήμασταν μαζί το 2012 μπορεί να πει ότι υπήρχαν τρεις πυλώνες εποπτεία, εξυγίανση, εγγύηση καταθέσεων με την, εν, έννοια της αλληλεγγύης που δεν μπορούμε να λυσμόνουμε αυτό ήδη από το 2012 αναφερόταν ένα Άλλο στοιχείο για να ολοκληρωθεί το ευρώ είναι η προοδευτική ολοκλήρωση ενός γνήσιου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου με δημοκρατικό έλεγχο που μπορεί να καταστεί ευρωπαϊκός θεσμός και όχι καθαρά διακυβερνητικός μηχανισμός όπως είναι τώρα. Και η Ευρωζώνη και η διακυβέρνηση της που πολλοί ανέφεραν ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι για να έχουμε ένα γνήσιο εργαλείο σύγκλησης και μείωσης των ανισοτήτων. Η δημοκρατική διακυβέρνηση ταυτόχρονα με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι μια άλλη προϋπόθεση. Αποφάσεις που λαμβάνονται σε, κλειστούς, ε, σε κλειστά αίθουσε χωρίς δημοκρατικό έλεγχο δεν είναι το ίδιο καλές με αυτές που λαμβάνονται με δημοκρατικό έλεγχο. Γι' αυτό και πρέπει το Eurogroup, αποτελεσματικό βέβαια μέσον και εργαλείο, να υφίσταται, να εκτίθεται στο δημοκρατικό έλεγχο. Δεν μπορούμε αυτή τη διάσταση να τη λησμονήσουμε. Ένα τρίτο ζήτημα για να καταλήξω, λαϊκισμός που ο κύριος Μπόρκη παραδείγματι ανέφερε. Και θέλω να πω εδώ ότι οι λαϊκιστές δεν είναι εχθροί. Συνήθως και αυτό συμβαίνει αντίστροφα από την άλλη πλευρά. Όταν βλέπει κανείς έναν εχθρό προσπαθεί να τον υποτιμήσει, να τον αποδιαρθρώσει, να τον κατηγορήσει με ψευδείς συνήσεις, ειδήσει. Αυτό μπορεί να συμβαίνει από ορισμένε πλευρές, όχι από εμά. Αντιθέτως βέβαια αν συμβαίνει ε, να υπάρχει ρατσισμός, αντισημιτισμός κτλ. Βεβαίως και τον καταδικάζουμε και εκεί βλέπουμε τον εχθρό σε αυτού του τύπου την συμπεριφορά του. Την άλλη εκδοχή που είναι ο λαϊκισμός την βλέπουμε σαν αντίπαλο, ναι, που πρέπει όμως και να αντικρούσουμε, όχι να, ε, να καταστρέψουμε. Η Ιταλία, παραδείγματι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η παρουσία της Ιταλίας μέσα στη ζώνη του ευρώ. Κύριε Μπον, και εσείς είπατε πρόσφατα, γράψατε μάλλον, ότι αν δεν μπορέσει να αλλάξει η Ευρώπη με το αποτέλεσμα των προσεχών ευρωεκλογών, θα πρέπει να βγει η Ιταλία από αυτήν. Ε, νομίζω ότι ακριβώς εκεί είναι το μεγάλο σας λάθος και εκεί θα κάνουν την επιλογή οι Ευρωπαίοι και οι Ιταλοί. Θα μείνουν μέσα στην Ευρώπη, θα μείνουν στην Ευρωζώνη για να τη βελτιώσουν. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει το μεταρρυθμιστή από τον λαϊκιστή, ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι εντοπισμός, ο εντοπισμός των προβλημάτων, των ε, ανεπαρκειών, η φιλοδοξία στην επίτευξη των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και η υπεράσπιση του ευρώ ως ε, επιτυχημένης ιστορίας είναι πράγματα που συμφιλιώνονται, δεν είναι πράγματα αντιφατικά μεταξύ τους. Πολλά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Μπόργκη θα πρέπει να αξιολογηθούν και να συγκριθούν με το ποια θα ήταν η κατάσταση χωρίς το ευρώ. Νομίζω ότι θα ήταν χειρότερη η κατάσταση χωρίς το ευρώ, όχι καλύτερη. Άρα μπορεί κανείς ταυτόχρονα να υπερασπιστεί το ευρώ και να το γιορτάσει, γιατί είναι πράγματι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για την ανάκαμψη Τη οικονομική και νομισματική κυριαρχία σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και μπορεί από την άλλη να κάνει κριτική ανάλυση. Και εγώ στην ομιλία μου άσκησα κριτική στα χρόνια της λιτότητας και ε, εντοπίσα τα προβλήματα, ότι το τωρινό οικοδόμημα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λύσει τα προβλήματα στο σύνολό τους. Έχουμε ορίσει μια φιλόδοξη πολιτική ατζέντα που είναι κοινά τα στοιχεία της, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, βελτίωση των εργαλείων για τη διαχείριση των κρίσεων, ε, δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων από πλευράς δημοσιονομικών και προϋπολογισμού για να έχουμε ανθεκτικότητα, σταθεροποίηση και ε, δυνατότητα ανάκαμψης και βεβαίως πλήρη συμπερίληψη του κοινωνικού πυλώνα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ενίσχυση των επενδυτικών μας δυνατοτήτων γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές και αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων που θα πρέπει να είναι πιο αντικυκλική και λιγότερο προκυκλική. Λέγοντας όλα αυτά, συγχαίουμε διαφορετικές φάσεις. Εγώ δεν νομίζω ότι από το 2011 μέχρι το 2014 είχαμε λιτότητα και ασφαλμένη οικονομική πολιτική. Αμφισβητώ όμως και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτή την ε, δημοσιονομική σταθερότητα και ε, ε, με ε, αυτή την πληθωριστική και επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκείνα τα χρόνια, για όλα αυτά τα χρόνια. Χρειαζόμαστε κοινά εργαλεία. Άρα ισχυρότερο προϋπολογισμό και σύστημα ίδιων πόρων για τη χρηματοδότηση αυτού. Ιδαλλιώ ε, είμαστε σε παιχνίδι μηδενικού αθρίσματο. Είτε κόβουμε την πολιτική συνοχή γιατί θέλουμε να πρημοδοτήσουμε κάποια άλλη, είτε κόβουμε από κάπου αλλού και δεν έχουμε ε, ε, αποτελέσματα. Η φιλοδοξία του 1,3% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη και συμφωνούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις για τους ίδιους πόρους και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, έτσι ώστε με αυτά τα έσοδα να χρηματοδοτηθεί ο προϋπολογισμός. Είναι απαραίτητο αυτό για να έχουμε αποτελεσματικές κοινέ πολιτικές. Είμαστε στα μισά της διαδρομής λοιπόν, έχουμε πετύχει πολλά και κανείς δεν αμφισβητεί τα σημαντικά αποτελέσματα που έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια χάρη στην ενωτική δυνατότητα δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι ένα από τα στοιχεία του ενεργητικού μας τα πολύ σημαντικά. Με τις διαφορές που έχουμε θα πρέπει να ε, συμπορευτούμε και να υιοθετήσουμε μια φιλόδοξη πολιτική ατζέντα. Αυτό μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια για να είναι πιο επικοδοματική η συζήτηση για την πορεία που θα ακολουθήσουμε και για να πείσουμε περισσότερο τους εκλογείς εν ώψη των επόμενων ευρωεκλογών. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, από πλευράς της Ρουμανικής Αντιπροσωπείας, θα ήθελα να εκφράσω τις βαθιές μας ευχαριστίες, να σας πω ότι είμαστε ευγνώμονες, διότι ήρθατε εδώ και μαριαστήκατε μαζί μας ιδέες, προτάσεις, σκέψεις για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Ε, ευχαριστούμε γιατί σχολιάσατε τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε και που αντιμετωπίζουμε. Όμως είναι ημέρα εορτασμού. 20 χρόνια έχουν περάσει, μεγάλος ο δρόμος και δύσκολος. Ας είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες στους προκατόχους μας που δημιούργησαν αυτό το μοναδικό εργαλείο ε, και πρέπει να κάνουμε κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δώσουμε και εμείς τη σκητάλη με επιτυχία στην επόμενη γενιά. Σας ε, περιμένουμε με χαρά στο Βουκουρέστι ε, για να ε, συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Now we

Ista, ne?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 No, nema ne pa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

No, sam je, sam je u pisku demo se priznat ne, da je u širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik, ne. Ja, da pač kateri popustijo potem, ne, razumem. To je, tak je, ne, pač. Ma ne, sej ni bistveno.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

pa kar ni grozno na obrazu, ne res tega ne moraš čakati, ukazati, da ti ne bomo več ne moreš narediti sam data Ja, nimaš A ja, ja. Moje ona, Μερού, με συνήθιζε ο Άσεπα. Ήταν je podoban. Ne boš to hnatančen.

Ο Σίκα. Ο Σίκο, ο διφύ, ο Σίκο, ο πασχοφάιου, ο κ. Νέκο. Α, η Αναφάμουστο, ο διφύ. Ο διφύ. Ναι, διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ο διφύ. Ναι, ναι, ναι.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

morning Καλημέρα σας. Κύριε Γιάνκου της Ρουμανικής Βουλής, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητέ Πρόεδρε Γκουαλτιέρη, χαίρομαι, είναι μεγάλη τιμή για μένα που σας βλέπω εδώ, στην 8η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδα Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διακοινοβουλευτική εκδήλωση που υποδέχεται το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο και σήμερα έχουμε 123 ε, μέλη, 123 βουλευτές από 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 5 υποψήφιες χώρες και από την Ουρβηγία και την ε, Ελβετία. Ε, μία από τις κύριες προτεραιότητες μου ως, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να ε, φέρουμε την ευρωπαϊκή πολιτική και τα θεσμικά της όργανα πιο κοντά στους πολίτες. Τα εθνικά κοινοβούλια δραματίζουν κέριο λόγο για την επιτεύξη του στόχου αυτού. Πρέπει να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη και την, ε, ε, την προσήλωση των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κοινή στόχοι μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ένα νέο όρομα για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις για την αναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν για να το επιτύχει αυτό πρέπει να ενισχύσει, θέλει να ενισχύσει τη διακοινοβουλευτική συνεργασία. Και επιτρέψτε μου τώρα να συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα, την Ιταλική. Αυτές τις μέρες συζητούμε την ε, σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμείνου, την αποτελεσματικότητα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών μας, της ε, σταθερότητας, της ανάπτυξης, της διακυβέρνησης της οικονομίας. Η εκτιμήση για το 2019 που μας παρουσίασε πριν από μερικές ημέρες η Ευρώπη δείχνει μια επιβράδυνση για την Ευρώπη, ύστερα από μερικά χρόνια κατά τη ε, οποία είχε επιτρέψει μέχρι και 14, 14 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας να ανακτηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε την επανάληψη στην Ήπειρό μα τη ύφεση που είχαμε πριν από 10 περίπου χρόνια. Προσωπικώ ανησυχώ ιδιαίτερω γιατί είναι πολύ σημαντικέ και οι ανισότητε οι περιφερειακέ αλλά και οι κοινωνικέ που παραμένουν στην Ευρώπη μα. Ε, υπάρχουν ορισμένε περιφέρειες που έχουν επιβράδυνση, ήδη βλέπουν την ύφεση στον ορίζοντα και έχουν ε, ποσοστά ανεργίας που ξεπερνούν και το 10%. Η ανεργία των νέων είναι στο απαράδεκτο επίπεδο του 42,3%. 42,3% στην Ελλάδα, 34,1% στην Ισπανία, 32,6% στην Ιταλία. Στην ένωσή μα, το 10% των νέων ούτε σπουδάζει ούτε εργάζεται. 120 εκατομμύρια ένα στους τέσσερις δηλαδή Ευρωπαίοι κινδυνεύουν από την φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η τεχνολογική επαν, ε, επανάσταση, η τεχνολογικη επανασταση κυκλοφορία των κεφαλαίων και των αγορών μπόρεσαν να επιτρέψουν ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα ε, ε, δημιούργησαν και ε, έναν αγώνα δρόμου προς τα κάτω ως προς τις συνθήκες ε, της απασχόλησης, τις φορολογικές αλλά και τις περιβαλλοντικές. Οι μεταναστευτικές ροές ανεξέλεγκτες πολλές φορές και η χαμηλού κόστου, το χαμηλού κόστου εργατικό δυναμικό, έφερε πολύ μεγάλε δυσκολίε ε, για τι πιο αδύναμες ε, κλάσεις, για τις πιο αδύναμες τάξεις των κοινωνιών μα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια αποφασιστική απάντηση, να δείξουμε ότι η Ευρώπη ενωμένη, πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική μπορεί να δώσει τι απαντήσεις στα προβλήματα αυτά. Μόνο μαζί μπορούμε να δώσουμε μια αποτελεσματική απάντηση στι μεγάλε παγκόσμιες προκλήσει ε, που προέρχονται από τι ΗΠΑ, την Κίνα, τη Ρωσία ή την Ινδία. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανάπτυξη που θα φέρει και θέσει εργασία αλλά και ευημερία για όλου του Ευρωπαίου. Το ε, δικό μα μοντέλο τη κοινωνική οικονομία και αγορά είναι αυτό που πρέπει να προστατέψουμε. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τι βασικέ αξίε, τη ελευθερία, τη αξιοπρέπεια του ανθρώπου πρέπει να ξεκινήσει μια βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη, μια βιομηχανική πολιτική με επενδύσεις, με έρευνα, με καινοτομία, ε, υποδομές, πιο δίκαιο εμπόριο και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει συγκεκριμένα μέτρα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που θα πρέπει να ενσωματωθούν στο προσεχή προϋπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε υποστηρίξει την αύξηση μέχρι 120 εκατομμυρίων του προσεχούς κοινωνικού ταμείου, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση με τι ενεργού πολιτικέ τη υποστηρίξη ε, για την απασχόληση των νέων και για την μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασία. 5,5 δισεκατομμύρια επίση το Ταμείο InvestEU επενδύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων προγράμματα για την ψηφιακή Ευρώπη, την έρευνα, τα περιφερειακά ταμεία, την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και τα μεγάλα δίκτυα των υποδομών και ε, δεν φτάνουν ακόμα και αυτές οι επενδύσεις δεν αρκούν. Χρειάζονται νέες τεχνολογίες προς ε, εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων δεν μπορούν να είναι, από, δεν μπορούν να είναι οι γίγαντες του web ε, ε, σε θέση να επιβάλλουν τους όρους τους εργαζόμενους ή στα φορολογικά, στη διαφάνεια, στην προστασία της ε, δημόσιας, του ιδιωτικού βίου και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο για τις σημαντικές συμφωνίες που έχουν να κάνουν και με την οδικία για το δικαιώματα του πνευματικού δημιουργού, τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής που επιτρέπει πιο δημιουργική Ευρώπη, αλλά και ένα χώρο δικαίου για τους μουσικούς μας, τους ηθοποιούς, τους συγγραφείς, τους δημοσιογράφους, ε, τους συγγραφείς και έτσι μπορούμε να έχουμε ε, νέες προτάσεις για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανταγωνιστική στον κόσμο με τον ορίζοντα Ευρώπη που φτάνει με αύξηση του 5% στα 120 δισεκατομμύρια όπως προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και του κοινωνικού αισθού και συγκρατεί τον κοινωνικό αισθό της Ευρώπης. Έχουμε στήσει λοιπόν την εισαγωγή ιδιαίτερων κεφαλαίων σε πολλά προγράμματα υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στις μεγάλες ευρωπαϊκές υποδομές και στο πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, για την άμυνα αλλά και για το διάστημα. Πρέπει να αναπτύξουμε όλο το δυναμικό της ενιαίας αγοράς, ξεκινώντας από τις υπηρεσίες, την ενέργεια, το, η ψηφιακή οικονομία πρέπει να συμπληρωθεί η ευρωπαϊκή αγορά με τη δημιουργία θέσεων εργασία, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δικαιωμάτων των καταναλωτών για να προσεγγίσουν και οι λιγότερο ανεπτυγμένε περιφέρειε, αυτέ που είναι πιο προηγμένε και πλούσιε. Με την έκθεση για τη στρατηγική για την ενιαία αγορά που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, προχωρούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Η ιστορική μα αγορά θα πρέπει να εξασφαλίσει και περισσότερη δικαιοσύνη και, δημοσιονομική, και φορολογική δικαιοσύνη και αρμονία συγγνώμη, δεν μπορούμε να έχουμε φορολογικούς παραδείσους ή μηδενικά επίπεδα φορολόγησης. σε ανάπτυξη και η δικαιοσύνη ολοκληρώνουν έτσι την αγορά των κεφαλαίων, την Τραπεζική Ένωση, αλλά και την ε, Δημοσιονομική, Οικονομική και Πολιτική Ένωση. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινό νόμισμα χωρίς να μιλούμε για πιο ομοιογενή επίπεδα ανταγωνιστικότητας και για καλύτερη οικονομική και κοινωνική σύγκληση. Βεβαίω, καλό είναι και το νέο μέσο για τη σταθεροποίηση των επενδύσεων και η πρόταση για την εγκαθίδρυση ενό κοινού νομισματικού ταμείου, Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου που θα προσφέρει μέσα υποστήριξη και μετά των μεταρρυθμίσεων και αντιμετώπιση των προβλημάτων και των κρίσεων. Θέλουμε αυτό το ταμείο όμω να συμπεριλαμβάνεται μέσα στου μηχανισμού Ευρώπη για να έχει μια διακυβέρνηση οικονομική πολύ πιο διαφανή και δημοκρατική. Πιστεύω ότι και το Ευρωπαϊκό όπω και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν πολύ περισσότερο στι διαδικασίε λήψεων αποφάσεων και μέσω μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού, των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημερινή συνάντηση. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε και να δώσουμε απάντηση στου προβληματισμού των πολιτών, ξεκινώντα από την καταπολέμηση ενεργεία των νέων, τη παράτυπη μετανάστευση, με τα εργαλεία τη ασφάλεια και τη άμυνα, αντιμετωπίζοντα και την ε, κλιματική αλλαγή στα γαλλικά και με τα συμπεράσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από του αρχηγού κυβερνήσεων να. Ε, τοποθετηθούν ε, στο μέλλον της Ευρώπης. Τους προσκαλούμε λοιπόν στις ολομέλειές του μας ε, και ε, με τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους εμπλουτίζουμε τη συζήτηση με τρόπο ανοιχτό και διαφανή. Μια συζήτηση η οποία επιτρέπει και στο Ευρωπαϊκό αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια να συμβάλλει και να ενισχύει τη δημοκρατική διαδικασία της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχύσει έτσι την νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την τελευταία δεκαετία τα κόμματα τα ευρωπαϊκά που συνεισέφεραν στην ε, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση διπλησίασαν ε, τις ψήφους τους. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έδειχναν εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Γεωγραφικές ε, περιοχές που είχαν χαμηλή απασχόληση Εκεί είναι που ψηφίζει ο κόσμος κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Κυρίως στον τομέα των οικονομικών ε, πολιτικών ε, και να ενισχύσουμε την ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κοινοβουλευτική εβδομάδα θα συνεισφέρει στην υπευθυνότητα της διακυβέρνησης της οικονομικής στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτό που ήρθατε εδώ αυτή τη βδομάδα. Καρποφόρες εργασίες σε όλους.